Καλησπέρα σας. Περιμέναμε λίγα λεπτά προκειμένου να αρπάξουμε λίγα ακόμα μέλη, αλλά κάποιοι έχουν παραμένει στον τρίλογο. Δεν θα καθυστερήσουν πολύ, φαντάζομαι. Τέλος πάντων, με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τον κύριο Ταβάρες, Κάλλος Ταβάρες, πρόεδρο της Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών. της ΣΕΖΡ. Φαντάζομαι ότι χαίρονται και εκείνοι ιδιαίτεροι που, ιδιαίτερα που καταλήξαμε σε συμφωνία για την ε, οδηγία IFM. Και η τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν το Δεκέμβριο του 2009 για μια ανταλλαγή απόψεων. Ενώ τώρα η σημερινή μα συζήτηση είναι μέρο τακτικών ανταλλαγών απόψεων που έχουμε με την, μεταξύ κοινοβουλευτικών επιτροπών και επιτροπών επίπεδου του επίπεδου 3. Βεβαίως θα αλλάξουν όλα αυτά όταν ε, θεσπιστούν και νέες αρχές και ελπίζουμε να δούμε πολλούς εκπροσώπους τους. Τώρα ο κύριος Σταβάρης θα μας κάνει μια παρουσίαση για τις πρόσφατες δραστηριότητες της ΣΕΖΑΡ και επίσης όλες τις ε, πρωτοβουλίες της Επιτροπής οι οποίες θα ασχοληθούμε με τον αρχιτεκτόνημα της χρηματοπιστωτική εποπτεία που θα αρχίσει να ισχύει από τον Ιανουάριο του 2011. Υπάρχουν πολλές νομοθετικέ προτάσεις οι οποίες θα δώσουν ιδιαίτερε αρμοδιότητες σε αυτές τις ευρωπαϊκές αρχές. Μετά την παρουσίαση του κ. Ταβάρες θα έχουμε προφανώς συζήτηση με τα μέλη τη Επιτροπής. Σα ευχαριστώ για τον λόγο. Καλησπέρα σας Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών. Όμως η Επιτροπή αυτή ήδη στα πλαίσια του υπολόγου της λογοδοσίας που τη διέπει έχει συζητήσει πολλές φορές με το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον να σας δώσουμε μια ενημέρωση για τι δραστηριότητε μας το τελευταίο εξάμεινο. Εγώ θα σας παρουσιάσω μια επισκόπηση ουσιαστικά της πρόσφατης εκθεσής μας και βεβαίως και τα προσωπικά μου σχόλια θα ήθελα οπωσδήποτε να κάνω κατά τη διάρκεια αυτής της παρουσίασης, τα οποία είναι πιο πολύ μακροπρόθεσμα και διορατικά, παρά αφορούν το πρόσφατο παρελθόν. Προκειμένου να έχουμε μετά και μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Θα ξεκινήσω ε, παρουσιάζοντας την άποψή μου για τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει από την συνεχιζόμενη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Θα τα συνοψίσω σε τρεις πτυχές. Πρώτα απ' όλα η ανάγκη να καλυφθούν τα ρυθμιστικά κενά με εποπτεία και παρακολούθηση όλων των αγορών και των οικονομικών παραγόγων για τις οικονομικές οντότητες και τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους. όπως για τα θέματα για τα οποία πρόσφατα επιτέχθη συμφωνία, Πρόεδρε, και χαίρομαι ιδιαίτερα που συνέβη αυτό σε επίπεδο θεσμικών οργάνων. Έπειτα, η διαφάνεια πρέπει να παράσχουμε στους επενδυτές ε, όλες τις δυνατότητες καθώς και στις ρυθμιστικές αρχές όλες τις δυνατότητες για να επιβάλλουν τους κανόνες τους. Έπειτα, κατά τρίτον, οι συστημικοί κίνδυνοι δεν θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζονται ως ένα ζήτημα που αφορά μόνο τις τράπεζες, τον τραπεζικό τομέα, αλλά και την αγορά των κινητών αξιών, όλες τις δομές και τα χρηματοπιστωτικά οικονομικά ιδρύματα. Αυτές τις ανάγκες τις ε, διεπίστωσε πρόσφατα και η Επιτροπή για το, και το Συμβούλιο για τον Ευρωπαϊκό Συστημικό Κίνδυνο. Θα ήθελα λοιπόν να εντοπίσω κάποια σημεία που προκύπτουν από την εξέταση της Γιώσκο ότι υπάρχουν παράγοντε του συστημικού κινδυνού που μπορούν να περιλαμβάνουν κάποια μοτίβα συμπεριφορά διανομή ε, ε, κάπου από συνθήκε ε, πίεση για ορισμένα επενδυτικά προϊόντα. Ε, Επίση, κάποιε διακοπέ στην αγορά ή δυσκολίε στην κενά στην ακαιρεότητα της αγοράς. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση να αντιμετωπιστούν σε ευρύ επίπεδο οι μη επαρκείς επενδύσεις, η μη επιβολή των ρυθμιστικών κανόνων, οι ανεπάρκειες των απαιτήσεων διαφάνειας και ούτω καθεξής. Επιπλέον, στην ίδια κατεύθυνση, θα πρέπει να έχουμε μια συμμετρική αντίληψη της ε, οικονομικής σταθερότητας. Θα πρέπει σε αυτή να βασιστούμε. Δηλαδή, υπερβολικά αυξανόμενες τιμές μπορεί να ζημιώσουν και να αποσταθεροποιήσουν τις ήδη σε ύφεση αγορές και οι ρυθμιστές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία και να δράσουν αναλόγως σε όλες τις περιπτώσεις. Εδώ έχουμε έναν τομέα που έχει αφιερώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Επιτροπή μας, η ΣΥΖΑΡ, ε, ενισχύοντας το έργο της τον τομέα τη οικονομικής ανάλυσης, καθώς και στην αξιολόγηση του κινδύνου, τι τάσει και τα ευάλωτα σημεία των ευρωπαϊκών οικονομικών και χρηματοπιστωτικών αγορών. Τα πορίσματα συστηματικά ε, μεταβιβάζονται στην FSC και στην EFC και δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά τον περασμένο Ιούλιο. Του τελευταίου μήνε επίση συνεργαστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τι άλλε επιτροπέ του επίπεδου 3 προκειμένου να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική λειτουργία του ESRB από την 1η Ιανουαρίου και μετά. Προχωρώντα τώρα από τα διδάγματα του παρελθόντο στι αναγκαίε μεταρρυθμίσει. Κεντρικό στόχο θα πρέπει να είναι να διασφαλίσουμε ασφαλέστερε αγορέ και υποδομέ. Μία βασική μεταρρύθμιση εδώ αφορά τι αγορέ των ε, κινητών αξιών, OTC, ε, όπου ένα μέρος της κρίσης μεταβιβάστηκε και μεταδόθηκε πρόσφατα. Οι πρόσφατες επιτροπέ, ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την αγορά των παραγόγων καταδεικνύουν τη σωστή κατεύθυνση για τις μεταρρυθμίσεις. Όμως πιστεύω ότι θα πρέπει οι αρχές αυτές, OTC, να παραταθούν και να καλέκουν και τις αγορές των παραγόγων. Έτσι θα αναχαιτήσουμε τις τρευλώσεις της αγοράς, τις, παρα... τις ε, καταχρήσεις της αγοράς και την κερδοσκοπία. Επίσης έχουμε και τις πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, την, ε, για το short selling και τα credit default swaps. Ε, εδώ χρειάζεται τεχνική συμβολή η οποία προσφέρθηκε από τη ΣΥΖΑΡ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προχώρησε στην υιοθέτηση του κανονισμού ΕΜΙΡ, κάτι που είναι μια ισόρροπη βάση για μεταγενέστερες ε, ε, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Η παγκόσμια αγορά δείχνει ότι η τελική πρόβλεψη νομοθεσίας δεν μπορεί να αγνοεί τις αντίστοιχε, τους αντίστοιχους κανόνες που ισχύουν σε άλλα νομοθετικά συστήματα, κυρίως λόγω των διασυνδέσεων μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Εδώ ο νόμος Dodd-Frank ε, καταδεικνύει την ίδια κατεύθυνση με αυτή του σχεδίου κανονισμού της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης για την αγορά παραγωγών OTC. Ωστόσο υπάρχουν διαφορές στην ε, νομική δομή, στο περιεχόμενο και στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προκειμένου να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για την ρυθμιστική διαιτησία. Παραδείγματα απόκλησης στο λεπτομερές περιεχόμενο των κανόνων Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ μπορούν να εντοπιστούν και στο πεδίο, δηλαδή το φάσμα των παραγόγων που είναι επιλέξιμα για την ε, υποχρεωτική καθάριση μέσω του CCP και τον ορισμό των ε, υποχρεώσεων εκαθάρισης. Εδώ η οργάνωση και η διεξαγωγή των ε, δραστηριοτήτων CCP ε, περιλαμβάνουν απαιτήσει για την ε, πώληση και ορίζουν συγκεκριμένα περιθώρια. Όμως οι ρυθμιστές, η CFTC και η CEC, έχουν πρωταρχικό εδώ ρόλο στην ανάπτυξη μιας διοργανωτικής και επιχειρηματικής συμπεριφοράς σε σχέση με τα πρότυπα της CCP. Η νομική αυτή δομή είναι πλήρως ε, ενσωματωμένη στην Αμερικανική νομοθεσία, ενώ στην Ευρώπη κάποια στοιχεία λείπουν. Ιδίως ε, στα θέματα διαφάνεια και εμπορίου. Αυτό θα μα απασχολήσει κατά την αναθεώρηση MIFID. Αυτέ οι δύο νομοθετικέ διαδικασίε δυστυχώ δεν συνέπεσαν χρονικά. Η αναθεώρηση MIFID και το σχέδιό τη πρόκειται να δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2011. Ενώ στι Ηνωμένες οι αρχέ εποπτεία και οι ρυθμιστικέ αρχέ, η CFTC και η CEC, e έχουν ήδη περάσει στη φάση υλοποίηση τη ρυθμιστική βάση που προβλέπεται από τον νόμο των Frank. Προκειμένου να διασφαλίσουμε και τη ρυθμιστική σύγκληση και έναν ενεργό ρόλο για την Ευρώπη στη, στη διαμόρφωση συγγνώμη, της υλοποίησης είναι, ε, είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι ρυθμιστές, η ΣΥΖΑΡ και η ΕΣΜΑ, καθώς και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκινήσουν εξ αρχής έναν εντατικό διάλογο ε, με τις Αμερικανικές αρχές και μεταξύ τους. Η ΣΥΖΑΡ ήδη έχει ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία σε συνεργασία με την, μέσω μάλλον τη CFTC και τη CSE. Επίση, ενδείκνεται στι συγκεκριμένε περιπτώσει να διατηρήσουμε την απαραίτητη ευελιξία στην νομοθετική δραστηριότητα. Πράγματι, αυτή είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με την ε, ρύθμιση σε αυτόν τον τομέα. Από την άλλη, το θέμα αυτό είναι ε, εξαιρετικά τεχνικού χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντε στην αγορά έχουν αποδείξει ότι είναι ταχύτατοι στην ανταπόκρισή του στι νέε κανόνε και δημιουργούν νέε προκλήσει προ του ρυθμιστέ. Υπ' αυτέ τι συνθήκε, ένα σημαντικό μέρο τη ρύθμιση θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να υλοποιηθεί μέσο μέσω υποχρεωτικών τεχνικών προτύπων, τα οποία να σχεδιαστούν και να αναθεωρηθούν από την άσμα, ΕΣΜΑ. Αυτή είναι και η προσέγγιση που έχουν θετήσει οι Αμερικανικέ Αρχέ, οι οποίε έχουν αφήσει πολλέ αρμοδιότητε στη CFTC και την CEC. Ιδίω ό,τι αφορά του τεχνικού ορισμού και τι λύσεις που προτείνονται. Σε αυτό το σκηνικό, σε αυτό το πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση του ΕΜΕΡ και τη ΜΥΦΙΔ, των αναθεωρήσεών του δηλαδή, είναι καθοριστική σημασία. Υπό τι παρούσε συνθήκε, η εξελισσόμενη αναθεώρηση ΜΥΦΙΔ δεν είναι απλώ μια κλασική αναθεώρηση. Θα πρέπει να περάσουμε σε μεταρρύθμιση επί τη ουσία, πιστεύω, που να ενσωματώνει και τα διδάγματα που έχουμε αποκομίσει, από το πρόσφατο παρελθόν. Τολμώ εδώ να υποδείξω τι πιστεύω ότι είναι οι 7 αρετέ που θα πρέπει να διέπουν την αναθεώρηση Μίθιντ. Πρώτα απ' όλα να διασφαλίσουμε υλοποίηση του consolidated tape όπως ονομάζεται, της ε, συνολικής ενημερώσεως για τις αγορές, έπειτα να διευρύνουμε το πεδίο υποβολής εκθέσεων για τις συναλλαγές, έπειτα να έχουμε τις καλύτερες αρχές εκτέλεσης που να, να είναι αποτελεσματικές, έπειτα υποχρεώσεις διαφάνειας που να ισχύουν για όλα τα εργαλεία και τις αγορές, έπειτα να εφαρμόσουμε νέες ε, διαδικασίες για τις συναλλαγές, όπως τις συναλλαγές ψηλής συχνότητας, Έπειτα, όποτε είναι δυνατόν τα ομόλογα και τα παράγωγα OTC να περάσουν σε οργανωμένους ε, σε οργανωμένα εμπορικά κέντρα και έπειτα να δοθούν ευκαιρίες ε, για να μειωθεί η ρυθμιστική απόκληση μεταξύ των κρατών μελών. Έπειτα ε, πιστεύω ότι η ΕΣΜΑ θα έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει εδώ στο να υιοθετήσουμε ένα ενιαίο σύνολο κανόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τους επενδυτές και να διασφαλίσουμε διαφάνεια για όλες τις αγορές ε, και αυτό θα είναι σπονδυλική στήλη οποιασδήποτε αναθεώρησης μύθη και όλων των σχετικών μεταρρυθμίσεων. Εδώ υπάρχει μια αυξανόμενη τάση να διανέμονται περιπλόκα προϊόντα σε, σε αγοραστές ε, σε επίπεδο λιανικής πώλησης. Γι' αυτό λοιπόν απαιτείται η ενίσχυση και η περαιτέρω αποσαφήνιση των κανόνων MIFID για την προστασία των επενδυτών και πρέπει να υπάρχει και ένα πεδίο ίσων ευκαιριών για τα ε, χρηματοπιστωτικά προϊόντα ελληνικής πώληση στο μέλλον. Ε, στο μέλλον επίσης οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, ιδίω η ΕΣΜΑ και βάσει του άρθρου 6α θα πρέπει να ε, φροντίζει για την επαρκή υλοποίηση. Η ΣΥΖΑΡ έχει δώσει τεχνικές συμβουλές σε πολλούς τομείς της αναθεώρησης MIFID και η Task Force 3L3 έχει ετοιμάσει πρόσφατα μία σχετική έκθεση. Στην τελευταία συζήτηση της Task Force, της ομάδας δράσης, συζητήθηκαν οι δυνατότητες δράσης για το θέμα της λιανοποίησης, όπως, όπως ονομάζεται, utilization των περίπλοκων προϊόντων, ε, τα οποία έχουν πάρει διάφορες μορφές, usage, ETN, MTN και ούτω καθεξής, καθώς και την υλοποίηση του άρθρου 6α του κανονισμού ΕΣΜΑ. Η ανάγκη να παρακολουθήσουμε τις επιπτώσεις από τα διδάγματα του παρελθόντος είναι σημαντική και για το παρόν. Ε, έχουμε τους ε, φορείς βαθμολόγησης, ο σχετικός κανονισμός βρίσκεται στην τελική του φάση και η ΣΥΖΑ έχει εκδιπλώσει πλήρω τι λειτουργίε τη στη μεταπατική περίοδο, φροντίζοντα οι απαραίτητε προετοιμασίε για την ΕΣΜΑ να έχουν ε, προσδώσει τι απαραίτητε αρμοδιότητε που προβλέπει ο κανονισμό που ακόμη συζητιέται. Η πραγματική και επιδόσεις ε, των εποπτικών λειτουργιών της ΕΣΜΑ πρέπει να εξασφαλιστούν ώστε να υπάρχει και κατάλληλη επιβολή αυτών των μέτρων. Ωστόσο θέλω να υπογραμμίσω ότι προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί ο κανονισμός θα πρέπει να συμπληρωθεί με μέτρα που ασχολούνται με το πρότυπο θεμελίωση του CRA και το να αποφύγουμε την υπερβολική εμπιστοσύνη στις βαθμολογίες αυτές ε, κυρίως με την ε, υιοθέτηση των βαθμολογιών αυτών από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θα πρέπει να προβλέψουμε και τις συγκρούσεις συμφερόντων. Ε, η πρόληψη σε κάθε περίπτωση είναι προτιμότερη από την εποπτεία και την αντιμετώπιση των ε, δυσκολίων εκ των υστέρων. Εδώ επίσης ένα άλλο σημαντικό βήμα είναι να καλυφθούν τα αριθμιστικά κενά, αυξάνοντας το φάσμα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που καλύπτονται. Αυτό είναι σημαντικό για σκοπούς διαφάνειας. Στην διάρθρωση της υλοποίησης σε όλες τις νομοθεσίες, οι κανόνες και τα πρότυπα θα πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αμοιβαιότητα η ΕΣΜΑ μπορεί να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά της, όπως τα αποδίδουν οι νέοι κανονισμοί. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο των ρυθμιστικών ευθυνών της ΕΣΜΑ σε τομείς όπου δεν έχει την ανάλογη πείρα, χωρίς να της ε, αποδώσουμε το ανάλογο οικονομικό τους ανάλογους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους ε, όπως δηλώνονται στους πρόσφατα σχέδια και προτάσεις προπολογισμού. Τα τελευταία μου λόγια θέλω να τα αφιερώσω στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, ιδίως στην ΕΣΜΑ. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο κανονισμός για τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές δεν είναι σίγουρα η άριστη μετάφραση στην πράξη των προτάσεων Λαροζιέρ. Ντέλα ε, για παράδειγμα, έκδοση υποχρεωτικών τεχνικών ε, προτύπων ε, με την απέτηση να υιοθετούνται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι που εννοεί ότι θα πρέπει να βασίζονται, υπονοεί ότι θα πρέπει να βασίζονται στην συνθήκη. Ε, οι ρυθμιστικέ αρχέ επίση που προσδίδονται στην ΕΣΜΑ θα μπορούσαν να είναι πιο φιλόδοξε. Ε, οι αρμοδιότητε που προσδίδονται στην ΕΣΜΑ είναι μεν σοβαρέ και σε τομεί που δεν είναι τόσο πολύ γνωστοί, όπω οι αγορέ OTC, το short selling, ή ε, Φορεί ε, βαθμολογία και οι εναλλακτικέ επενδύσει. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι η αναθεώρηση των οδηγιών MIFID MAD και τη διαφάνεια, θα ενισχύσουν τον ρόλο τη ΕΣΜΑ και τη δυνατότητά τη να πετύχει ένα, σύνολο, ένα ενιαίο σύνολο κανόνων. Το να κάνουμε αυτό που οφείλουμε βάσει των ε, σημερινών προοπτικών δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι η ΕΣΜΑ θα αναλάβει όλε τι αρμοδιότητε που ήδη έχουν προβλεφθεί για το ρόλο τη και θα τι ασκήσει αποτελεσματικά. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα τεράστιο έργο που πρέπει να επιτελεστεί και αν πρόκειται να συμβούν όλα αυτά, μπορούμε να αναμένουμε σε μια μελλοντική αναθεώρηση η ΕΣΜΑ να αποκτήσει περαιτέρω εξουσίες ε, που προκύπτουν από τη δίδυση στο καθεστώς. Τώρα, το, αν, το να συνεχίσουμε απλώ να παραπονιόμαστε ή το να μην είμαστε επαρκεί στην άσκηση των καθηκόντων μα, σημαίνει ότι δεν θα πάρουμε περισσότερα στο μέλλον. Πιστεύω πραγματικά ότι η ΕΣΜΑ θα διαμορφωθεί ανάλογα με τι επιθυμίε των μελών τη. Αυτό βεβαίω εξαρτάται και από τα άτομα, αλλά και από το ρόλο που θα διανοματίσει ο πρόεδρο στο να διασφαλίσει ισχυρή δράση για αυτή την αρχή. Είναι σημαντικό και το Συμβούλιο των Εποπτών να ασκήσει πραγματικέ εξουσίε όπω τι προβλέπει το καθεστώ τη ΕΣΜΑ. Από την άλλη, διαδικασία για την έγκριση υποχρεωτικών τεχνικών προτύπων θα απαιτεί ανοιχτό και διαρκή συντονισμό μεταξύ των φορέων της αρχής και των υπευθύνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το λέω εγώ αυτό ως πρόεδρος της ΕΖΑΡ και ενθαρρύνοντας αυτό το είδος το συντονισμό στη διάρκεια του διαστήματο που έχω αναλάβει τα καθήκοντά μου. είναι τεράστιε λοιπόν οι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε, από κάθε άποψη και ιδίω ω προ τι προσδοκίε των επενδυτών. Είμαστε υποχρεωμένοι να τι καλύψουμε τι προσδοκίε αυτέ και πρέπει να είμαστε στι ρυθμίσει μα αποτελεσματικοί, ευέλικτοι και ε, εύστοχοι. Θα πρέπει οι αγορέ να λάβουμε υπόψη ότι εξελίσσονται διαρκώ, οι κανονισμοί αλλάζουν και η ΕΣΜΑ μπορεί να συμβάλλει τα μάλα στο να έχουμε την απαραίτητη ρυθμιστική απόκριση. Πιστεύω λοιπόν ότι πλέον βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Είναι πολλά αυτά που έχουμε ήδη επιτύχει, αλλά και πολλά αυτά που απομένουν να γίνουν. Αυτά που έχουμε μπροστά μας να κάνουμε βέβαια είναι πολύ σοβαρά και για να μην πω και πολύ πιο κατεπήγοντα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει ένας κατάλογος ομιλητών. and Peter, I've now got... Και ο Σβέν, όλα, Φειό, ποιος άλλος, Σαϊάν, η Ελίζα, Ούντο Κέι, Πίτερ, Μάρκος, όλοι όσοι άκουσαν το όνομά τους. Έχουμε 20 λεπτά. Ποιος άλλος ε, θέλει. Δύο λεπτά ο κάθε ομιλητής. Προτείνω να κάνουμε ομάδες ε, τεσσάρων ερωτήσεων, αλλά πραγματικά θα πρέπει να περιορίσετε το χρόνο ομιλίας σας. Ο Ούντο. Κύριε Ταμπάρες, θα ήθελα να σας πω, καταρχήν καλωσορίσατε εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας και η πρώτη εντύπωση που μας κάνατε μπαίνοντα είναι πραγματικά αν θέλετε μία εντύπωση που δεν ήταν σωστή γιατί ουσιαστικά είμαστε υπέρ της εργασίας σας, των προσπαθειών σας και σας στηρίζουμε. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Μιλήσατε για τις απειλές, μιλήσατε για τους κινδύνους των αγορών. Όσον αφορά τη ρύθμιση των hedge funds, έχουμε πετύχει μία ενιαία στάση. Δεν ξέρουμε όμως όσον αφορά τις προθεσμίες υλοποίησης, αν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλα αυτά πριν το ξεκίνημα της νέας μεγάλης κρίσης. Πείτε μας λοιπόν, εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα και ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι, οι μεγαλύτερες πηγές κινδύνων. Και δεύτερο, ακριβώς επειδή μιλήσατε και για τη ρύθμιση των αγορών OTC, ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά το πολύ κρίσιμο θέμα της αξιολόγησης για την κερδοσκοπία στα, στις πρώτες ύλε και στα ίδια διατροφής. Σήμερα ξέρουμε ποιες είναι οι προτάσεις της ε, Επιτροπής, η οποία πραγματικά διστάζει. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Um, I'd like to come to, uh, Ευχαριστώ και εγώ θα κάνω την ε, ερώτηση όσον αφορά το προσωπικό το οποίο θα προσληφθεί για την ΕΣΜΑ και θα αρχίσει να εργάζεται τον Ιανουάριο. Υψηλού επίπεδου προσωπικό και βάσει όλων των ρυθμίσεων, των κανονισμών και των οδηγιών που αφορούν την ΕΣΜΑ, Ξέρουμε σήμερα ποιος είναι ο ρόλος ε, αυτού του οργανισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τις, την εκαθάριση και όλους τους άλλους τομείς. Πιστεύετε ότι τα 80 άτομα που προβλέπονται αρκούν γιατί γνωρίζετε την υπάρχουσα εργασία σας και την επιπλέον φαντάζομαι μπορείτε να την αξιολογήσετε. Το προσωπικό λοιπόν που θα προσληφθεί προσλαμβάνεται βάσει των τεχνικών τους γνώσεων της εμπειρογνωμοσύνης τους και βεβαίως υπάρχουν πολλές ε, ρυθμιστικές αρχές σε επίπεδο εθνικών ε, αρχών. Τα κράτη δηλαδή προσφέρουν αυτή την εμπειρογνωμοσύνη. Αυτοί θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με την ΕΣΜΑ. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Κοιτάξτε, κάνετε πάρα πολύ περίπλοκες ερωτήσεις και υπάρχουν μόνο 30 δευτερόλεπτα για απάντηση. Όσον αφορά την κρίση, η εκτίμηση των κινδύνων και των απειλών είχαν γίνει με πάρα πολύ επιπόλαιο τρόπο, θα έλεγα είχαν ε, εκτιμηθεί οι πραγματικοί κίνδυνοι και δεν υπήρχαν τα απαραίτητα αποθέματα. Τι μπορούμε λοιπόν να πούμε από εδώ και πέρα. Χρειαζόμαστε νέους κανόνες, χρειαζόμαστε νέους κανόνες οι οποίοι να αρχίσουν να ε, ισχύουν ε, γρήγορα και βεβαίως χρειαζόμαστε και υψηλότερη ρευστότητα από αυτή που υπήρχε και βεβαίως ε, κεφάλαια σε υψηλό επίπεδο για αποθεματικό και ως collateral. Αυτό βεβαίως απαιτεί μία διαδικασία απόφασης πάρα πολύ γρήγορη. Σήμερα ξέρουμε όλοι ότι τα πρότυπα των ΗΠΑ διαφέρουν από αυτά τη Ευρώπη. Τι θα κάνουμε για να υπάρξει εναρμόνιση. Σας ευχαριστώ. Εσείς ασχοληθήκατε και με το flashcraft στη Νέα Υόρκη και σαφώς υπάρχουν σήμερα τρόποι για να εξουδετερωθεί η επόμενη κρίση με συγκεκριμένες φόρμουλες. Έγιναν οι τέσσερις ερωτήσεις, αλλά έχετε μόνο τέσσερα λεπτά για να απαντήσετε. Έχετε το λόγο, κύριε Ταβάρες. So, as, as quickly... Uh, uh, ναι, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η βασική κίνδυνη για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κατ' με, είναι ότι δεν θα πρέπει θα πρέπει να υιοθετήσουμε μεταρρυθμίσει το συντομότερο δυνατόν. Όπως σα εξήγησα, υπάρχουν πολλοί τομεί ε, του χρηματοπιστωτικού τομέα και ως προ τα προϊόντα και ως προ τα τραπεζοπιστωτικά ιδρύματα που δεν ρυθμίζονταν αρκετά. παρά το γεγονό ότι η κρίση ξεκίνησε από το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ, εξαπλώθηκε σχεδόν σε όλες τις αγοράς και σε όλα τα χρηματοπιστωτικά συστήματα. Και επομένω τώρα θα πρέπει να τους δώσουμε τα κατάλληλα μέσα για να εποπτεύσουν και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ζητήσουμε στου στους ε, ε, να είναι υπόλογοι σε κάποιον. Προ το παρόν δεν υπάρχουν αυτά τα εργαλεία και θα θυμάστε και την ε, πράξη για, τη μελλοντική, για το μελλοντικό εξυγχρονισμό που υιοθετήθηκε το 2000 που δεν περιλάμβανε τίποτα και δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε μέσα για την εποπτεία και για να έχουμε μια εικόνα για το τι γίνεται με τις αγορές ομολόγων και παραγόγων, συμπεριλαμβανομένων και των αγορών ε, οι οποίες ε, ε, αποτέλεσαν και αντικείμενο συζήτησης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν περάσει ήδη τρία χρόνια από την κρίση και ουσιαστικά είμαστε στο ίδιο νομοθετικό παρελθόν, περιβάλλον όπως ήμασταν και στο παρελθόν. Επομένως είναι κατεπήγον να δώσουμε τα μέσα στους επόπτες ώστε να έχουν τη δυνατότητα ε, να ε, εργαστούν το συντομότερο δυνατόν. Και αυτό φυσικά ισχύει και για τα αγαθά και για τις ε, αγορές τροφίμων διότι οι αγορέ παραγόγων σχετίζονται και με τα αγαθά και το πρόβλημα είναι πανομοιότυπο. Πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη ρύθμιση και να δώσουμε στι νομοθέτες τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Για το πολύ σημαντικό θέμα της πρόληψης προσωπικού, πράγματι έχουν δοθεί πολλές επιπλέον εξουσίες ε, για τη λειτουργία του CASR. Ε, καταρχάς, ε, οι τεχνικές προδιογραφές αλλάζουν τελείως τη λογική και τη μεθοδολογία της αρχής, αλλά όπως ε, σας είπα και στην αρχική μου παρέμβαση, μας δίνονται και εξουσίες σε τομείς οι οποίοι δεν ρυθμίζονταν στο παρελθόν, που είναι τελείως καινούργοι και είναι πολύ τεχνικά ε, τα σημεία αυτά και οι γνώσεις μας προς το παρόν βρίσκονται από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της αγοράς. Επομένως, η πρόσληψη προσωπικού θα πρέπει να γίνει κατά τρόπον ώστε να έχουμε άτομα με προσόντα, κατά πάσα πιθανότητα να προσλάβουμε και ανθρώπους της αγοράς που γνωρίζουν πολύ καλά αυτούς τους νέους ε, τομείς ε, παρέμβασης ε, της ESM και επίσης είναι εξίσου επίγον διότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας από 1η Ιανουαρίου αλλά θα πρέπει να υπάρχει και αρκετός χρόνος ώστε να προσλάβουμε τα κατάλληλα άτομα. Το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε χωρίς να έχουμε και τα κατάλληλα μέσα στη διάθεσή μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κάποια κατανόηση ως προς την ESM και να μην τη ζητήσουμε να λειτουργεί ε, πλήρως από 1η Ιανουαρίου. Εγώ και οι συνάδελφοί μου συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο περιθώριο ευελιξίας ε, για τον μελλοντικό πρόεδρο για να μπορέσει να ε, χειριστεί τα θέματα της μεσαίας διαχείρισης. Να επιλέξουμε τους κατάλληλους ανθρώπους και να μην κάνουμε μία αυτόματη μετάβαση της, ε, του Διοικητικού Συμβουλίου και της διαχείρισης του CSR στην ΕΣΜΑ. δεν έχει κανένας ε, το δικαίωμα να διατηρήσει τη θέση του στην ε, CESR. Επίσης, ε, στο μέσο επίπεδο χρειαζόμαστε επιπλέον ανθρώπους, κατά πάσα πιθανότητα χρειαζόμαστε και καλύτερους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τα καλύτερα δυνατά άτομα για να ασχοληθούν ακριβώς με αυτά τα θέματα τα οποία είναι τόσο τεχνικά. τι μπορούμε να κάνουμε και τι κάνουμε ήδη από τώρα. Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία εξέτασης ε, του συνολικού οργανογράμματος ε, του ΡΙΣΕΣΜΑ βάσει των νέων καθηκόντων που αναλαμβάνει, αλλά βέβαια η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από τον ε, μελλοντικό πρόεδρο και από τον μελλοντικό διευθυντή, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα θα αναλάβουν καθήκοντα το Μάρτιο του 2011. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε λίγο υπομονετικοί να λειτουργήσουμε γρήγορα μεν, αλλά ε, να λειτουργούν και τα πράγματα σωστά από την αρχή. Τώρα, ως προς τους δυνητικούς κανόνες ε, για τις ε, κεφαλαϊκές απαιτήσεις, νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντική γιατί πρέπει να έχουμε διατήρηση της σταθερότητας και όπως σας είπα και στην αρχική μου παρέμβαση αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο τις τράπεζες τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά πρέπει να έχουμε και ασφάλεια και στις αγορές, στις υποδομές, επομένως ε, το να καθορίσουμε κατάλληλα επίπεδα κεφαλαίου για το CCP ή για οποιαδήποτε άλλη υποδομή της αγοράς είναι πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε επίσης και νέους τομείς. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε συγκεκριμένη εμπειρία του παρελθόντος, διότι στις τράπεζες μπορεί κάποιος να εξετάσει τι έγινε στο παρελθόν, να δει τι πήγε στραβά και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Αλλά στους τομείς αυτούς ε, ουσιαστικά ε, προχωράμε στα τυφλά. Ξεκινάμε από το μηδέν και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά και πάλι με τα κατάλληλα άτομα, αλλά και με τη δέουσα ευελιξία. Επειδή ακριβώς πρόκειται για νέους τομείς, ε, ε, κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξουν σφάλματα στην αρχή. Δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση να τα κάνουμε όλα σωστά από την αρχή. Ε, γι' αυτό ακριβώς προτείνω να δοθεί μεγάλη ε, βελιξία στα δεσμευτικά, στις δεσμευτικές τεχνικές προδιαγραφές της ΕΣΜΑ και να μην έχουμε πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Διότι αν έχουμε πάρα πολλέ λεπτομέρειε στο βασικό κανονισμό, θα είναι πάρα πολλά ε, δύσκολο να τα διορθώσουμε στο μέλλον και όπω σα είπα, είναι πολύ τεχνικά αυτά τα θέματα. Για το flash crash, ε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο στι ΗΠΑ να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη με το flash crash. Δυστυχώ, πρόκειται για ένα ε, flash crash το οποίο διέρχεσε πάρα πολύ λίγο, Ελάχιστε ώρε και διορθώθηκε αμέσω, επομένω δεν υπήρχαν ε, συστημικές επιπτώσεις. Όμως ε, και πάλι μπορεί κάποιο να συνάγει κάποια καλά συμπεράσματα, διότι πρέπει να εξετάσουμε αυτέ τι νέε μορφέ εμπορίου, να τις κατανοήσουμε καλά. Πρόκειται για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν πολύ καλά οι επόπτες και θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί εδώ και θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση όχι μόνο για να αποφεύγονται τέτοιοι κίνδυνοι, διότι μπορεί να είναι συστημική κίνδυνη εάν το flash crash διαρκούσε περισσότερο από, περισσότερο, από λίγες ώρες, αλλά αν αυτοί οι αλγόριθμοι έχουν ενσωματωμένους ε, αγο... Ε, τρόπους εκμετάλλευσης αγοράς ή οτιδήποτε άλλο. Δεν σας λέω ότι τα περιλαμβάνουν αυτά, αλλά θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν τα περιλαμβάνουν αυτά οι αλγόριθμοι. I'll take Peter, then Sven, then. Peter, Sven, Peter. Ευχαριστώ πολύ. Πόσα άτομα θα πάρετε στην Αρμόδια Επιτροπή, γιατί για μας είναι πολύ ύψιστη η προτεραιότητα αυτή. Πόσους θα βάλετε από την ΕΣΜΑ σε αυτήν την ειδική επιτροπή. Λιγότερο από δύο. Εξηγήστε μας γιατί σε αυτή την περίπτωση. Αν είναι λιγότερο από τα δύο τα άτομα που θα διορίσετε, να μας πείτε γιατί παρακαλώ. Ο Σβέν. Καταρχήν καλωσορίσατε. Μεγάλη χαρά ήταν για μας ε, που επεξεργαστήκαμε και τον προϋπολογισμό σας αλλά και τις αρμοδιότητές σας. Καταρχήν θα ήθελα να σας ρωτήσω, από ό,τι ξέρω, εξετάζεται τις επιπτώσεις ε, των δραστηριοτήτων short selling και την ε, μείωση της βαθμολογίας ε, των κρατών από τους φορείς αξιολόγησης. Θέλετε να μου πείτε ποια είναι τα αποτελέσματα, ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε σε αυτήν τη δραστηριότητα. Και θα κάνω και την ίδια ερώτηση με τον Πίτερ αλλά για κάτι άλλο. Νέες αρμοδιότητες για την προστασία των καταναλωτών. Πόσα άτομα θα προσλάβετε, πόσα άτομα θεωρείτε ότι θα χρειαστούν για αυτήν την υπηρεσία, συγκρίνοντας βεβαίως με αυτό που συμβαίνει για παρόμοιες δραστηριότητες της Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ταβάρες, πιστεύετε ότι η CSR και οι ρυθμιστικές αρχές για 27 κράτη-μέλη, εάν υλοποιήσουν ε, τις υποχρεώσεις τους και διαπιστώσουν προβλήματα στις χρηματαγορές, θα μπορούν ε, να προτείνουν μέτρα για να μετριαστούν τα προβλήματα. Το 2005 η CSR πρότεινε σε μια ομάδα εργασίας την ανάλυση της δραστηριότητας των οργανισμών αξιολόγησης. Και σαν αποτέλεσμα τότε, το 2005, δεν βγήκε απολύτως κανένα αποτέλεσμα από αυτήν την αξιολόγηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πόσα άτομα στην Μικτή Επιτροπή. Πρόκειται ακόμα για θέματα που τα συζητούμε. Πάντως όχι λιγότερο από δύο. Όχι λιγότερο από δύο, σίγουρα. Για το ξεκίνημα τουλάχιστον. Θα ξεκινήσουμε με δύο. Πολύ συγκεκριμένα. Καταλαβαίνετε ότι η Μικτή Επιτροπή ακόμα είναι υποσυζήτηση με τις επιτροπές που θα συνεργαστεί και ενδεχομένως θα ληφθεί και η απόφαση για τον αριθμό των μελών. Αλλά πραγματικά όχι δεν θα είναι λιγότερο από δύο άτομα. Παντώ στην ερώτησή σας. Και θα προσέξουμε πολύ αυτή τη μικρή επιστολή. Σας το λέω με σοβαρότητα. Τώρα, οι σχέσεις μεταξύ CSR νομίζω αναφερθήκατε κυρίως σε σχέσεις μεταξύ CBS για τη δραστηριότητα short selling. Κοιτάξτε, το εξετάζουμε ιδιαίτερα όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ ε, των τιμών του short selling στις ε, αγορές τους και των CDS. Στις 15 Δεκεμβρίου θα υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν θέλω τώρα να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Αλλά επειδή μιλήσατε και για το θέμα της ε, αξιολόγησης ε, των οργανισμών αξιολόγησης, της υποτίμησης, της ε, επιδείνωσης της βαθμολογίας. Αυτό που είναι γνωστό σήμερα είναι ότι αυτή η αξιολόγηση, αυτή η βαθμολογία θα πρέπει να πάψει να έχει τόσο σοβαρές επιπτώσεις, να γίνει άνευ σημασίας. Και αυτό θα γίνει μόνο και εφόσον οι κυβερνήσεις ε, δημιουργήσουν μεγαλύτερη διαφάνεια. Εάν υπάρχει πλήρης διαφάνεια για το τι κάνει η κυβέρνηση και αν τα λεγόμενα μιας κυβέρνησης και τα στοιχεία που δημοσιεύει είναι αξιόπιστα και ορθά, Καταλαβαίνετε ότι η αξιολόγηση αυτών των οργανισμών πραγματικά δεν θα έχει τόση σημασία. Παίζει ρόλο λοιπόν εδώ να δούμε τι πληροφορίες δίνουν οι κυβερνήσεις τους επενδυτές. Η άλλη ερώτηση για την προστασία των καταναλωτών είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα. Αυτό βεβαίως κοιτάμε την νέα ε, ρύθμιση. Ξεκινήσαμε με το άρθρο 6α και όπως είπα και στην παρουσίασή μου, ανησυχούμε ιδιαίτερα για την προοδευτική διανομή όλο και περισσότερων ε, περίπλοκων προϊόντων σε μεμονωμένους επενδυτές. Και στην τελευταία ολομέλεια μας, μια ομάδα υψηλού επίπεδου έχει αναλάβει το θέμα αυτό της προστασίας των καταναλωτών και το θέμα είναι πώς αυτό το άρθρο 6α θα πρέπει να υλοποιηθεί στην πράξη από την ΕΣΜΑ. Το ερώτημά σας λοιπόν, πόσα άτομα στην ΕΣΜΑ, δεν ξέρουμε ακριβώς τον τελικό αριθμό, βεβαίως, διότι πολλοί, αν θέλετε, θα πάρουν την απόφαση αυτή, κατά την άποψή μου. Πάντως, ο τομέας αυτός σίγουρα θα πρέπει να αποτελέσει ένα τομέα σημαντικής ε, δραστηριότητας για την ΕΣΜΑ. Ε, τελευταία ερώτηση. Έχετε δίκιο ότι το θέμα αυτό δεν ήταν θέμα αρμοδιότητας των ρυθμιστικών αρχών, αλλά βεβαίως έγινε τομέας αρμοδιότητας, καθότι δόθηκαν κάποιες αξιολογήσεις, βαθμολογίες σε κάποια προϊόντα που δεν ήταν αξιόπιστες. Θα αναλάβουμε λοιπόν πλήρως από εδώ και πέρα τις νέες μας αρμοδιότητες, συμπληρώνοντας την ρύθμιση και εξετάζοντας βεβαίως το ρόλο αυτών των ε, οργανισμών αξιολόγησης. Οι τρεις τελευταίοι ομιλητές, λέει η Πρόεδρος, παρακαλώ πολύ να κάνουν τις ερωτήσεις τους σύντομα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πώς βλέπετε το να υπάρχει μια, ένας ευρωπαϊκός φορέας βαθμολόγησης, ευρωπαϊκή εταιρεία βαθμολόγησης. Και αν πιστεύετε ότι ένας φόρος για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στη ρύθμιση των αγορών. Um, thank you. I wonder what... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το short selling. Το ECP λέγεται ότι οι ανώνυμες πληροφορίες για το short sale επαρκούν και πολλές πληροφορίες προς το ευρύ κοινό μπορεί να δημιουργήσουν επιζήμια συμπεριφορά. Ε, εξ όσων καταλαβαίνω, η CSR έχει διαφορετική άποψη. Μπορείτε να μας εξηγήσετε προς τι αυτή η διαφορά απόψεων. Thank you. Eh, Καλώ ήρθατε, δόκτωρα Ταβάρε, στο Κοινοβούλιο. Έχω δύο ερωτήσει. Ήδη τι έθιξαν προηγούμενοι συνάδελφοι. Παρ' όλα αυτά θέλω να επιμείνω. Πρώτον, το Κοινοβούλιο υπερασπίστηκε το να υπάρχει μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Αρχή και ψήφισε ανάλογο προπολογισμό. <clears throat> Ποιε είναι οι εναλλακτικέ που υπάρχουν τώρα, ώστε ήδη το Ιανουάριο να λειτουργεί με την ύψιστη δυνατή αποτελεσματικότητα αυτή η αρχή. Και έπειτα για τις credit rating agencies, τους οργανισμούς δανειοληπτικής ικανότητας. Εδώ λέτε ότι δεν θέλουμε να έχουμε over-reliance, υπερβολική εμπιστοσύνη σε, αυτές, σε αυτούς τους φορείς βαθμολόγηση. Όμως, για τα κρατικά χρέη, οι βαθμολογίες δεν παίζουν ρόλο. Θα ήθελα κάποια συγκεκριμένα σχόλια δυνατόν. Um, Ευχαριστώ. Για το θέμα των οργανισμών αξιολόγησης. Η ιδέα ενό ευρωπαϊκού οικοαξιολόγηση που ναι, μεν θα μπορούσε να έχει κάποια υπέρ, ε, είναι δύσκολη στην πρακτική εφαρμογή της ένας νέος οίκος αξιολόγησης θα πρέπει καταρχάς να γίνει αποδεκτός από τους χρήστες ε, των αξιολογήσεων και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μέχρι τώρα οι περισσότεροι χρήστες εμπιστεύονται τρεις οίκους. Το πιο σημαντικό δε είναι αυτό το οποίο είπα ήδη, ότι θα πρέπει να κάνουμε το παν προκειμένου να μην υπάρχει σύγκρουση συμφορέων και να υπάρχει άνοιγμα των αγορών. Και εκεί προκύπτει το ερώτημα. Αν μπορούμε να βρούμε ένα διαφορετικό τρόπο χρηματοδότησης των οργανισμών, ώστε οι αξιολογήσεις να μην ε, πληρώνονται από αυτούς που εκδίδουν τα προϊόντα, ε, ή τουλάχιστον να μην πληρώνουν το σύνολο της αξιολόγησης, ε, τότε θα, δεν θα έχουμε σύγκρουση συμφορώντων και θα μπορέσουμε να ανοίξουμε και την αγορά σε άλλους ε, φορείς, τους οποίους θα μπορούν να προσλαμβάνουν αυτοί που καταβάλουν ε, τα χρήματα. Αυτή είναι μια λύση την οποία θα πρέπει να συζητήσουμε. Δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ αυτό στο CSR, επομένως δεν θα επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να δούμε πρώτα τι γίνεται με τη σύγκρουση συμφορώντων και πώς μπορεί να πάψει να υφίσταται αυτή και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε την εξάρτηση. Ε, για παράδειγμα, ε, στον ε, ορισμό για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει ε, να υπάρχει να μην υπάρχει τόσο μεγάλη εξάρτηση από τις αξιολογήσεις. Αν μπορέσουμε να αναστρέψουμε αυτές τις παρενέργειες, θα ανοίξει η αγορά και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε και τη λύση σε αυτό το άνοιγμα, τουλάχιστον μερικώς. Για το θέμα του short selling. Ερίζουν οι απόψεις μεταξύ του ECP και του CESR. Καταρχάς ε, δεν θα έπρεπε να σας εκπλήσει ότι μπορεί να υπάρχει διάσταση απόψεων. Ε, ο δυνητικός ρυθμιστής δηλαδή να έχει διαφορετική άποψη από το ECSR είναι προκατάληψη και από τις δύο πλευρές. Ο καθένα το βλέπει από τη δική του σκοπιά ε, και θα πρέπει να το θεωρούμε φυσικό ότι υπάρχει διαφορετική άποψη. Οι κανόνε διαφάνειας που πρότεινε το CSR και που έχει αναλάβει δεχτεί το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα υπάρχει διαφορά, διότι ο τρόπος με τον οποίο αποκαλύπτονται οι θέσει του short ε, είναι ανώνυμες, ε, είναι συνολικά ποσά, επομένως είναι σημαντικό ή μάλλον εξίσου σημαντικό ε, όσο είναι η αποκάλυψη το γεγονός ότι λαμβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια τους, κίνδυνους, τους κινδύνους ε, για το next short selling, το πώς δίνονται οι παραγγελίες, ε, τι κανόνες προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά είναι ουσιαστικά ένας τρόπος ε, ρύθμισης του short selling που ελαχιστοποιεί τους κινδύνους τουλάχιστον αυτούς τους κινδύνους που μπορεί να έχει το short selling. η δημιουργία αυτής της νέας Ευρωπαϊκής Αρχής. Όπως σας είπα και στην αρχή, θα πρέπει να είναι μια ισχυρή αρχή που θα έχει και εξουσίες και αρμοδιότητες, τις οποίες θα πρέπει να ασκεί καταλήλως. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για να δημιουργήσουμε αυτή τη νέα αρχή, να προσλάβουμε τα κατάλληλα άτομα, να συνεργαστούμε μαζί τους και να καθορίσουμε και την, ε, τον οργανωτική δομή. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να ξεκινήσουμε ε, της εργασίας μας από την 1η της 2 Ιανουαρίου. Όπως σας είπα όμως, ε, όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν βαθμιδών. Ε, διότι ο νέος πρόεδρος και ο νέος εκτελεστικός διευθυντής θα αναλάμβουν καθήκοντα το Μάρτιο κατά πάσα πιθανότητα. Και αυτή η νέα αρχή θα πρέπει να έχει κάποιες σταθερές βάσεις. Γι' αυτό άλλωστε λέω πάντα ότι πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλο προπολογισμό, ε, να υπάρχουν κατάλληλοι οικονομικοί πόροι, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που μας ζητάτε, αλλά για το πρώτο χρόνο θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σόφρονες και να μην ζητάμε τα πάντα από την πρώτη στιγμή. γνωρίζουμε άλλωστε ότι κάποια στιγμή μέσα στο 2011 θα έχουν όλα ξεκινήσει να λειτουργούν και θα έχουμε και τα κατάλληλα άτομα στην κατάλληλη θέση. Όπως σας έλεγα υπάρχουν νέα καθήκοντα και νέες λειτουργίες, πολλές μάλιστα, Και γι' αυτό ακριβώ έχουμε επιστήσει και την προσοχή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και του είπαμε ότι χρειαζόμαστε και τα κατάλληλα μέσα για να κάνουμε αυτό που μα ζητάτε. Και φυσικά εννοείται ότι από εκεί και πέρα είμαστε υπόλογοι σε εσά για όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε που δεν είχαμε περισσότερο χρόνο να ολοκληρώσουμε περαιτέρω αυτήν ανταλλαγή απόψεων, αλλά βλέπετε τι συμβαίνει συνήθω. Τόσα μέλη τη Επιτροπή πόσο ενδιαφέρονται για το έργο σα. Πάντως σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις ε, τροπολογίες για τα credit rating agencies, για τους οργανισμούς δανειοληπτικής ικανότητας. Πάντως ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε και άλλη ανταλλαγή απόψεων μαζί σας ή μέσα τον ίδιο ή με κάποιον άλλον υπεύθυνο της ε, δικής σας αρχής. Θα προχωρήσουμε με τις, ψηφοφορίε με τις ψηφοφορίες εντός λεπτών. Μπορείτε να χειροκροτήσετε. Right, everybody, do you, do you have voting cards? Λοιπόν, έχετε όλοι τις κάρτες ψηφοφορίας σας. Εάν τις έχετε, βάλτε τις στο μηχάνημα. Εάν δεν τις έχετε, αρχίστε να πανικοβάλλεστε. Ο κύριος Φέγιο δεν έχει την κάρτα του. Υπερβάνς, ούτε και εκείνη. Okay, well, we'll, we'll, we'll worry about that θα ανησυχήσουμε όταν έρθει η ώρα. Για να κάνουμε μια δοκιμή. Άρχεται η ψηφοφορία. Όποιος είναι υπέρ, ας πατήσει το συν. Εγώ έχω γρήπη και είμαι ακόμα υπέρ. Λοιπόν, ε, δύο μόνο, εφτά μάλλον είναι χαρούμενοι και απέχουν, δύο δεν ξέρουν. Πρόεδρε, είπατε το πράσινο είναι το χρώμα της χαράς. Το κόκκινο δεν μας είπατε τι είναι. Μήπως είναι το πολύ χαρούμενο. Okay, we'll have another check. Okay, you can press anything you like then. Πατήστε ό,τι σας αρέσει. <laughs> A button that is. <laughs> Για κουμπιά μιλούσα. Look, be careful. This is being web streamed. Να προσέχουμε γιατί περνάμε και στο ίντερνετ. Right, okay, the vote's closed. We have to add that one. Right, we've got three, three, we've... Λήξη. Έχουμε μια κάρτα που δεν λειτουργεί λοιπόν. Βάλτε και μια τρίτη που δεν λειτουργεί. Ωραία. Έχουμε μια κάρτα λοιπόν πράσινη που δεν λειτουργεί. Έχουμε και μια κάρτα του ΕΛΚ που δεν λειτουργεί ή απουσιάζει. Λείπει για μια κάρτα των σοσιαλιστών. Ας ελπίσουμε να μην χρειαστούμε πολλές επαληθεύσεις. Τέλο πάντων κάποιο είναι στην Ινδία και εγώ έπρεπε να είμαι, αλλά τελικά δεν τα κατάφερα. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίε. Έκθεση για την ε, ετήσια έκθεση του, της, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του 2009. που έλεγε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Δεκα... Κατά μέρη, κατά τμήματα για τη 14, ψηφοφορία, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά κάποια χέρια δεν σηκώθηκαν καλά. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική σι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ή e. ε, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Επόμενη, σελίδα παράγραφος 5α νέο. Προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική για την παράγραφο 6α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε πάμε στη συμβιβαστική F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 εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο για την παράγραφο 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ σε δύο τμήματα μάλλον. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεν μπορώ να πω. Πρέπει να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πρόεδρε, ως έξυπνο ξέχασα την κάρτα μου. Τέσσερι λοιπόν. Εντάξει, θα το δούμε στο τέλος. Πολλοί σοσιαλιστές. Πάρα πολύ. Με τους σοσιαλιστές νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα, ψηφίζουν περισσότεροι. Λήξη. Θα ξαναρχίσουμε, θα ξαναψηφίσουμε, γιατί ψηφίζουν υπερβολικά πολύ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ξανά. Ωραία, πέρας. Πρέπει να προσθέσουμε και αυτούς που δεν ψήφισαν. Έχουμε έναν, δύο κατά. Ο κύριος Φόξ είναι κατά και ο κύριος Φέγιο το ίδιο. Και ένας υπέρ όμως δεν μετράει γιατί είναι δύο η κατά. Δεν εγκρίνεται λοιπόν. Συμβαστική I υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά δεν κρίνεται. Συγγνώμη, τα 44. Ποια είναι το πρόβλημα. 45. Στις 45 φτάσαμε. 45 υπέρ. Κατά αποχές δεν κρίνεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές δεν λέει πουθενά εάν καταπληκτεί. Δίκιο, είχα 47 και πάλι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52. Υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο παράγραφος 16 υπέρ. Πρέπει να ψηφίσουμε. Ναι, υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Δεκα... Συγγνώμη, 58 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 59 καταπίπτει. Διότι εγκρίθηκε η J. Συμβαστική K υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρι... απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. 64. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Ε, πέρας 37 ε, υπέρ Συγγνώμη, 19 υπέρ, 18 κατά. Κύριε Φέγιο, σας υπέρ ή κατά. κατά. Εσείς υπέρ. Και πάλι περνάει με μία ψήφο διαφορά. Ψηφίζουμε την 65 και την 66. Ωραία, 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική και α, υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική L υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική M υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 22 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 80 σε τρία τμήματα. Σωστά. 80 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά α το επαληθεύσουμε. Δεύτερο τμήμα. 80. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Απορρίπτεται. Ό,τι και αν κάνουν οι τρει που δεν έχουν κάρτα. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Μπορείτε να σκορδέτε τα χέρια παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 81. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφο 26. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική όμικρον. Ο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Παράγραφος 30. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θεολογικές σκέψει B και C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 7 να απελευθεύσουμε. 6 υπέρ λέει πρόεδρο, κατά αποχέ απορρίφθηκε νομίζω. Μάλλον είμαι πολύ γρήγορη. Ε. Θέλετε να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικώς. Α, έγινε. Εντάξει, να το ξανακάνουμε. Εγώ κοίταζα τα χέρια σας και εσείς ψηφίζατε με κάρτες. Σας παρακαλώ λοιπόν ψηφίστε πάλι. Τροπολογία 6. Ξαναψηφίζουμε. Πρέπει να υπολογίσουμε και τους τρεις χωρίς κάρτα. Ένας κατά ένα υπέρ. Είστε κατά. Είστε κατά. Δύο επιπλέον κατά. Είναι ίση η ψήφη. Άρα καταπέπτει. Πορύπτεται. Όχι, εκεί έχουμε ένα συν, ένα μείον εδώ και άλλα δύο μείον από εκεί. Είναι τρία τα πλήν. Τα προσθέτουμε λοιπόν 20 μείον 20. Άρα απορρίπτεται. Με 19 υπέρ. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίφθηκε. Συμβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική β, β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο με την ηλεκτρονική μέθοδο. Ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Ωραία. Τώρα πόσους θα προσθέσουμε. Έναν για τον κύριο Φέιο, έναν για τον κύριο Φόξ. 39 υπέρ. Και τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος. Και εσείς συν, και εσείς, και εσείς, άρα συν, τρία συν, άρα 38 προς 1. Κάποιος χάθηκε κάπου στον δρόμο. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. need a voting list. Voting list, No, sorry, here. So, granting... We're on to point 15. That's the one, yeah. Yep, okay. Right, is everybody ready? We're now moving on. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στην έκθεση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δέλτα, συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έψιλον, ε, υπέρ κατά. Συμβεβαστική έψιλον ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Τροπολογία 33 υπέρ Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Ένας κατά, ένας υπέρ και άλλο ένας υπέρ. Εγκρίνεται η τροπολογία 33. Ναι, εγκρίνεται ίσα. Συμβαστική F υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 36 ή 11. Α, όχι αποσυρθεί. 36. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές α, ε, εγκρίνεται. Συγγνώμη. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική, 18 ε, με προφορική, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική G, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 με προφορική υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η αρχική 19 χωρίς την προφορική, η αρχική 19 υπέρ κατά αποχές και αυτή απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και ψηφίνουμε ηλεκτρονικά το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί. Η επιπλέον, παρακαλώ πείτε μου πώς ψηφίζετε, συν, συν, συν. 37 υπέρ. Εγκρίνεται το κείμενο. Right, we now move on. Να περάσουμε τώρα στο σημείο υπέρθυνο 16 έκθεση του Hans Peter Martin για τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντοοικονομικούς λογαριασμούς. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Μπορούμε να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ, γιατί 15. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται, σαφώς, ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν οι άλλοι τρεις. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, πολλές αποχές. Να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 2, λοιπόν. τι γίνεται με τους επιπλέον που ψηφίζουν χωρίς κάρτα. Μήπως μπορούμε να την επαναλάβουμε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι όσοι έχουν κάρτα αυτή τη στιγμή. Πέρασε στις ψηφοφορίες λοιπόν. Απορρίπτεται λοιπόν, γιατί και με τις τρεις επιπλέον ψήφους πάλι δεν φτάνει η πλειοψηφία. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. τρία υπε σε τα τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να κάνουμε μια ηλεκτρονική παλήθευση αν θέλετε. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. 18-18. Τι ψηφίζουν αυτοί που δεν έχουν κάρτα. Απορρίπτεται λοιπόν. 16 υπέρ. Η 16 καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε το πρώτο τμήμα της 3. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται νομίζω. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ, κατά. Το ΕΛΚ δεν ψήφισε. Είστε υπέρ. Ωραία. Εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές Το ΕΛΚ μήπως μπορείς να μου πει αν είναι υπέρ ή κατά της 6. Ε, Είστε υπέρ, ωραία, εγκρίνεται τότε. Τροπολογία 23 υπέρ, με την προφορική τροπολογία 23 υπέρ κατά δεν ε, μπορώ να καταλάβω να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση για την προφορική τροπολογία της 23 ψήφισαν όλοι πέρασε της ψηφοφορίας εγκρίνεται Να περάσουμε στην τελική ψηφοφορία, θα γίνει ηλεκτρονικά. Η μία, δύο, τρεις επιπλέον ψήφοι. Ελήφθησαν υπόψη. 37 ψηφίσαντες. Συγχαρητήρια λοιπόν το στέκτη της νομοδότησης.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 colleagues, I, I apologize. Συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη, αλλά εγώ έχω γρήπη, γι' αυτό λοιπόν θα φύγω. Οι αντιπρόεδροι έχουν εξαφανιστεί όλοι, γι' αυτό την προεδρία θα αναλάβει η κυρία Λούλινγκ, η οποία θα έρθει εδώ να αναλάβει τα ενία. Συνήθως αυτό κάνουμε, ο γυρεότερος αναλαμβάνει. C'est pas la première fois. Hein. Déjà pendant les anciens. Και δεν είναι η πρώτη φορά που είμαι η αρχαιότερη. Και άλλες φορές στις προηγούμενες θητείες είχα αυτό το προνόμιο. Euh, euh, Περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Τροπολογίες της έκθεσης του κυρίου Γκοζές που αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης. Κύριε Γκοζές, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν είστε η πρεσβύτερη, είστε πρόεδρος. Βάλτε το μικρόφωνο σας. Λοιπόν, στην ημερήσια διάταξη έχουμε την εξέταση των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί από αρκετούς συναδέλφους, 100 τροπολογίες. Αυτό δείχνει ότι επικεντρωθήκαμε στα σημεία που θέλουμε να τροποποιήσουμε. Πρόκειται για ένα κανονισμό που υιοθετήθηκε το 2009 με σκοπό την εποπτεία από την ΕΣΜΑ. Μία έκθεση πρωτοβουλίας έχει ήδη αποφασιστεί. Ο συνάδελφος Βόλφης είναι εισηγητής. Και βεβαίως οτιδήποτε αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης, τα ελλείμματα των κρατών θα εξεταστούν σε αυτήν την έκθεση πρωτοβουλίας που θα αποτελέσει βάση για την Επιτροπή που θα υποβάλει κατόπιν το 2012 μία πρωτοβουλία, μάλλον το 2011 διορθώνει ο μιλητής, μία πρωτοβουλία ρύθμιση. το πρώτο εξάμεινο του 2011. Αύριο το πρωί θα συναντηθώ με τους σκιώδες εισηγητές για να προσπαθήσουμε να βρούμε συμβιβαστικές τροπολογίες σε κάποια από τα θέματα γνωρίζοντας ότι βεβαίως ε, ο χρόνος πιέζει. Στις 8 Νοεμβρίου θα γίνει μια δεύτερη συνάντηση για τις τροπολογίες, αν αυτό είναι απαραίτητο, και στις 9 θα συνεδριάσει η Επιτροπή μας, εδώ στις Βρυξέλλες. Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ, ο κ. Ρέντερς, ζήτησε η ρύθμιση, ε, ο κανονισμός συγγνώμη αυτός να εξεταστεί πριν το τέλος της προεδρίας του Βελγίου. Αυτό βεβαίως ε, χάρη στην επιτυχία της πρώτης ανάγνωσης. Τώρα, οι τροπολογίες στοχεύουν κυρίως το άρθρο 8α8β, πρόσβαση στην πληροφόρηση και το θέμα της διαφάνειας βεβαίως. Οι, τα αυτά προβλέπουν ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για τους οργανισμούς αυτούς και ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται με ε, εμπιστευτικό τρόπο, με δίκτυα δηλαδή που εγγυώνται την εχημήθεια ασφαλή δίκτυα. Οι οργανισμοί αυτοί οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να έχουν πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία ουσιαστικά αφορούν ούτε το 10, το 5% των ε, συναλλαγών και όπως λέει και ο κύριος Κλίνς, η έκθεση πρωτοβουλίας θα ασχοληθεί ευρύτερα με το θέμα αυτό. Άλλοι επιθυμούν όσον αφορά τα δομημένα χρηματοπιστωτικά εργαλεία να υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση για το κοινό στις πληροφορίες. Αυτό είναι ένα σχετικά λεπτό θέμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν πληροφορίες που παρόλο που πρέπει να υπάρχει διαφάνεια δεν θα πρέπει να είναι γνωστές στις αγορές. Απ' την άλλη υπάρχει και το επιχείρημα της ευρείας διάδοσης αυτών των πληροφοριών χωρίς να υπάρχει μία προνομιούχα πρόσβαση για τις ε, οργανισμούς αυτούς αξιολόγησης. Σήμερα υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος ε, χάρη στη μονοπωλιακή του θέση, στην ολογοπωλιακή του θέση έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και εδώ προτείνεται το άνοιγμα και η διεύρυνση αυτής της πρόσβασης. Όσον αφορά την ε, ΕΣΜΑ υπάρχουν οι τροπολογίες της κυρίας Μπόλς και του κυρίου Φόλς που προτείνουν να υπάρχει δυνατότητα έφεσης προσφυγής για να μπορούν να αποφευχθούν οι κυρώσεις. Οι κυρώσεις πάντως δεν θα πρέπει να επιβάλλονται από την ΕΣΜΑ. Προς το παρόν η Επιτροπή έλεγε ότι θα πρέπει να αποφευχθούν αυτές οι κυρώσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται Η ΕΣΜΑ θα είναι αυτή η οποία θα προτείνει τις κυρώσεις. Κάποιοι προτείνουν εδώ να πλαισιωθεί το ποσό των ε, κυρώσεων, έτσι ώστε να μην ξεπερνάει το 10% του ετήσιου ποσού των οργανισμών αξιολόγησης. Ο κύριος Κλίνς προτείνει η ΕΣΜΑ να κάνει μια ετήσια έκθεση η οποία θα υποβάλλεται στην Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά την αξιολόγηση του προσωπικού των αρμοδιοτήτων καθότι όλοι σήμερα αναρωτιόμαστε εάν το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτει η ΕΣΜΑ αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες αυτού του οργανισμού, καθότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί να υπάρχει διεύρυνση αυτών των αρμοδιοτήτων. Αυτά όσον αφορά τις τροπολογίες. Υπάρχει επίσης και το θέμα των μεταβατικών διατάξεων για το χρονικό διάστημα μεταξύ της αρχής της λειτουργίας της ΕΣΜΑ και της στιγμής που θα μπορέσει να υλοποιήσει τις αποστολές της. Και τέλος, υπάρχει και η έγκριση, η υιοθέτηση των οργανισμών αξιολόγησης που βρίσκονται σε τρίτες χώρες. Οργανισμοί αξιολόγησης που ακολουθούν διαφορετικούς κανόνες και τρόπο λειτουργίας από τις ευρωπαϊκές. Το θέμα αυτό ξεκίνησε όταν πήρε θέση το ΣΥΖΑΡ για την χρησιμοποίηση βαθμολογίας που προέρχεται από τρίτες χώρες. Και αν θυμάστε, συζητήθηκε έντονα το θέμα αυτό. Πώς δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε αξιολογήσεις που προέρχονται από τρίτες χώρες. Και αρχικά είχαμε πει ότι μόνο η αξιολόγηση οργανισμών που υπόκεινται στην ευρωπαϊκή ε, νομοθεσία θα λαμβάνονται υπόψη. Κατόπιν συζητήθηκε το θέμα και έγιναν δεκτές δύο εξαιρέσεις. Πρώτον, οργανισμοί που βρίσκονται σε χώρες που υπόκεινται σε ρύθμιση. Και μόνο και εφόσον υπάρχει μια συμφωνία εποπτείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αρχής, της ΕΣΜΑ δηλαδή, και της Αρχής Ρύθμισης και Εποπτείας της χώρας ε, με την οποία έχει συναυθεί η συμφωνία. Παράδειγμα, ο Καναδάς. Για βαθμολογίες που έχουν θεσπιστεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βαθμολογίες και αξιολογήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον έχει δοθεί πράσινο φως τις αξιολογήσεις αυτές από μία αρχή, από έναν οργανισμό, ο οποίος στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο, αυτή την αξιολόγηση και αυτή τη βαθμολογία βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων καθότι υπάρχει αυτή η ολιγοπολιακή κατάσταση στην αγορά αυτών των εποπτικών αρχών και των οργανισμών αξιολόγησης, έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι οργανισμοί που βρίσκονται σε τρίτες χώρες είναι θυγατρικές κάποιων οργανισμών που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη όλοι αυτοί οι κανόνες και ο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει βεβαίως περισσότερες ε, διευκρινήσεις για το θέμα αυτό. Η συζήτηση συνεχίζεται και επαναλαμβάνω ότι αύριο το πρωί θα συναντηθώ με τους και ηγητές για να συμφωνήσουμε όσον αφορά όλες τις τροπολογίες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Πολλά είναι τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όμως πρέπει να σας ενημερώσω κι εγώ από πλευράς φιλελευθέρων. Ο κύριος Κλίντς βρίσκεται στην Ινδία. Κυρία Μπόλς που θα τον αντικαθιστούσε σήμερα χρειάστηκε να αποσιάσει για λόγους υγείας. Η ομάδα λοιπόν Αλντέ μας ενημερώνει ότι η θέση της ομάδας θα παρουσιαστεί αύριο κατά την συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους σκιωδούς εισηγητές. Ο κύριος Πιτέλα, Εφόσον λείπει ο κύριος Κλίντς, ο κύριος Γίγκολτ, ο κύριος Φόξ, ο κύριος Κλούτ. Με συγχωρείτε, ο κύριος Φόξ. Ναι. Δεν αλλάξατε φίλο ακόμη. Κύριε Πιτέλα, έχετε το λόγο. Και όσοι συνάδελφοι θέλουν το λόγο, παρακαλώ να τον ζητήσουν. Κύριε Πιτέλα. Μα βλεπόμαστε συχνά στο Προεδρείο. Δεν μπορεί να με ξεχάσατε κύριε Λούλη και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Γκοζές ε, γνωρίζει ότι τον εκτιμώ και τον εμπιστεύομαι και συνεχίζω να τον εκτιμώ και να τον εμπιστεύομαι και για τον τρόπο με τον οποίο προχωρά αυτή την έκθεση. Τα σχόλια που έχω να κάνω αφορούν δύο άρθρα. Το άρθρο 8 το οποίο θέλει να ανοίξει περισσότερο τον τομέα της αξιολόγησης ε, ο οποίο από πλευρά μα θεωρείται ότι δεν έχει μεγάλο ανταγωνισμό και το άρθρο το οποίο αφορά τι κυρώσει. Όσον αφορά λοιπόν αυτά τα δύο προβλήματα, θα ήθελα να επαναλάβω τη θέση μου, την οποία είχα εκφράσει και κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και την οποία μετέφρασα και σε τροπολογίες. Πιο συγκεκριμένα, με τις τροπολογίες 106, 112, 114 και 115 ζητώ να δίνεται ε, εξουσία για τις κυρώσεις στην ΕΣΜΑ και όχι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί θεωρώ ότι καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της ενίσχυσης των νέων οργανισμών, των νέων αρχών, ώστε να μπορέσουν να διασφαλίσουν ότι θα γίνεται η αποτελεσματικότερη δυνατή εποπτεία. Ε, διότι αυτή τη στιγμή ε, την νομοθεσία δεν είναι δυνατόν να την αμφισβητούμε δημιουργήσαμε αυτές τις νέες αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνε για την εποπτεία και θα πρέπει να έχουν εξουσία. Τι σημασία έχει να έχει αυτή την εξουσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην την έχει η αρμόδια αρχή. Για να μπορέσει να υποστηριχθεί η πρόταση αυτή από νομική σκοπιά, προτείνω να υπάρχει ένα σαφή ορισμό για του περιορισμού για τι ε, κυρώσει και για το ε, φάσμα στο οποίο θα πρέπει να καθορίζονται οι κυρώσει. Αφενός θα πρέπει να δίνεται η εξουσία για τις κυρώσεις ε, στην ΕΣΠΑ, η οποία άλλωστε ε, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο. Θα ήταν παράδοξο για πρώτη φορά να συμφωνούμε σε κάτι εμείς και το Συμβούλιο και να μην συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τώρα το άρθρο 8, Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες ε, συναδέλφων που θέλουν να ενισχύσουν τη θέση που εκφράζει το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του εισηγητή Γκοζές και σε αυτές συμφωνώ κι εγώ και αυτό είναι και το πνεύμα της δικής μου τροπολογίας της υπαριθμών 68. Είμαι βέβαιο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα πρέπει να προχωρήσει στο θέμα των οίκων αξιολόγηση, ό,τι έκανε, ε, όπως έκανε και το 2009. Αν θυμάστε κύριε Γκοσέ, συνεργαστήκαμε πολύ καλά και θέλουμε να έχουμε μία σαφή και αυστηρή νομοθεσία. Απέτηση την οποία και εγώ νιώθω αλλά και άλλοι συνάδελφοι και αυτό το οποίο επιβεβαιώνει ίσως περισσότερο από όλα είναι οι τελευταίες ε, δηλώσεις του Προέδρου του Financial Stability Board, του, του Μάριο Ντράγκη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι στο επόμενο G20 θα παρουσιάσει κάποιες προτάσεις για το πώς θα πρέπει να μειωθεί η εξάρτηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης διότι τα αποτελέσματα ε, αυτής της αυτόματης διαδικασίας ήταν μάλλον απογοητευτικά. Εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Δράγκη και θα ήθελα να ζητήσω η Επιτροπή μας ε, και μετά το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια να επιβεβαιώσει αυτή την άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πιτέλα. Θέλετε κύριε Γκοζές να απαντήσετε αμέσως, ίσως είναι απλούστερο έτσι. Ή πρώτα να ακούσετε όλους τους και όδης Ας αφήσουμε όλους τους συναδελφούς να μιλήσουν, γιατί μπορεί να χρειαστεί και κάτι να προσθέσω. Ωραία. Κύριε Γκίγκολτ. Θα μιλήσω γερμανικά. Ήθελα να σχολιάσω ένα-δυο σημεία εδώ. Πρώτα απ' όλα, κάποιες από τις τροπολογίες του κυρίου Κλούτε, όπως τις βλέπω εγώ, θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί για την επόμενη έκθεση. Νομίζω προδικάζουν μια σημαντική συζήτηση που ακόμη δεν έχει γίνει. Είναι σαφές ότι υπάρχουν ζητήματα που δεν μπορούμε να τα λύσουμε τώρα. Ιδιαιτέρως, γιατί θα καθυστερήσουμε τις δραστηριότητες εποπτείας της ΕΣΜΑ και θα κολλησιεργήσουν και οι συζητήσει και στο Συμβούλιο και μεταξύ μα. Δεν θα είναι εύκολο να καταλήξουμε σε γρήγορη λύση. Υπάρχουν βεβαίω προτάσει που έχουν ως στόχο να επεξεργαστούν τη ρύθμιση της πρόσβασης στην αγορά. Δεν είμαι βέβαιος κατά πόσον η τροπολογία 42 λόγου χάρη είναι ορθή. Λέει ότι ένας ιδιώτης δεν μπορεί να δώσει τη γνώμη του για το καθεστώς ενός δημοκρατικού κράτους και την φερεγγιότητά του. Ό,τι άποψη και αν έχει ο καθένας, Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς τη συμμετοχή μικρών φορέων ακριβώς στην ε, αγορά. Είναι σαν να τους πετάμε έξω από το σύστημα και επειδή εδώ μιλάμε και για ανταγωνισμό, δεν είναι ιδεολογικό το θέμα, Το θέμα επί της αρχής, θα ήταν ενδιαφέρον να το συζητήσουμε πιο διεξοδικά. Υπάρχουν δύο τροπολογίες που ήθελα επίσης να σχολιάσω καθώ συζητάμε το ποιο πρέπει να λαμβάνει τι είδου πληροφορίε. Ναι, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Ιδίω, εξ όσων εγώ κατάλαβα, η Επιτροπή αυτή πάντοτε θα υπερμάχεται τη διαφάνεια. Είναι μια πάγια αρχή μα αυτή. Ουσιαστικά, αν θέλουμε να ανοίξουμε την αγορά δεν ε, μπορούμε να διαφωνήσουμε με την παροχή πληροφοριών για τους ε, οργανισμούς αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Αυτό λέει και η Επιτροπή όταν προτείνει το 10% των δομημένων προϊόντων να αξιολογούνται. Προφανώς αυτές οι πληροφορίες που να διατίθενται και στο κοινό. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι λογικό να εφαρμόζεται αυτό για τους μεγάλους μόνο οργανισμούς πιστοληπτική ικανότητα. Δεν πιστεύω ότι έτσι θα λειτουργήσει το σύστημα, ούτε, ούτε το κοινό πρέπει να αποκλειστεί από την όλη διαδικασία. Κάτι άλλο που θεωρώ σημαντικό είναι το ποια είναι η σχέση μεταξύ ΕΣΜΑ και εθνικών εποπτικών αρχών. Στο άρθρο 30 υπάρχουν εδώ κάποιες λεπτομέρειες. Νομίζω ότι αν θέλουμε να ακολουθήσουμε μια, μια ορθή εποπτική προσέγγιση, πρέπει να φροντίσουμε το προσεκτικά το τι αρμοδιότητε θα αναθέσουμε στην ΕΣΜΑ, Χωρί όμω να τις ε, αφαιρέσουμε πλαγίω και να τι αποδώσουμε σε εθνικέ αρχέ. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα όρια και ελπίζω να στηριχθούν οι τροπολογίε που υπέβαλα σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Αυτά έχω να πω προ στιγμή και πραγματικά ανυπομονώ για μια ενδιαφέρουσα και επικοδομητική πιστεύω συζήτηση που θα έχουμε και με τον Ζαμπόλ και με όλου του συναδέλφου αύριο το πρωί προκειμένου να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσει. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκόλτ. Ο κύριος Φόξ, Άσλι Φόξ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γκοτσέ για την δουλειά του σε σχέση με αυτή την έκθεση έω σήμερα και για την αυριανή συνάντηση που οργάνωσε. Είμαι σίγουρο ότι θα είναι επικοδομητική. Θα περιοριστώ στα άρθρα 8α και 8β την δημιουργία των ασφαλών ιστοτόπων. Διερωτώ με αν η Επιτροπή σκέφτηκε σοβαρά το τι ωφέλη πιστεύει θα προσθεθούν και τι κόστος θα έχουν τέτοια μέτρα. Διότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ένα παρόμοιο σύστημα. Και τα αποδεικτικά στοιχεία ως τώρα δείχνουν ότι δεν έχει ωφελήσει ιδιαίτερα. Επιβάλλει μάλιστα σοβαρότατο κόστος το σύστημα αυτό στην ε, δημιουργία κεφαλαίου, στις κέντρους κεφαλαίου. Εδώ δεν μιλάμε για τράπεζες ε, και καζίνο, αλλά μιλάμε για πραγματικές τράπεζες που απευθύνονται σε πραγματικούς ε, καταναλωτές, σε επιχειρήσεις. Και το κεφάλαιο τους ε, εξαρτάται από όλα αυτά, δηλαδή θα τους επιβάλλουμε υπέρμετρο κόστο ε, προκειμένου να διατηρούν τέτοιου ιστοτόπου για του οργανισμού πιστοληπτική ικανότητα. Δεν είναι το πρόβλημα του ίδιου, η ίδια, ο ίδιο ο ιστότοπο που θα προκαλέσει αυτό το κόστο, αλλά το ανθρώπινο δυναμικό ή το κόστο σε χρόνο. Το κάθε έγγραφο που θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο ιστότοπο θα πρέπει να περνάει από έναν ε, δικηγόρο. Εγώ στην ε, προηγούμενο, στον προηγούμενο επαγγελματικό μου βίο υπήρξα δικηγόρο και ξέρω ότι πρόσθετος φόρτος ε, σημαίνει αυτό για τους συναδέλφους μου. Ε, έτσι λοιπόν οι οργανισμοί πιστοληπτικής ικανότητας δεν θα περιλαμβάνουν τίποτα στον ιστοτόπο που δεν έχει ελεγχθεί νομικώς. Αυτό θα καθυστερεί όμως πάρα πολύ την διαδικασία συγκέντρωσης κεφαλαίου. Και αυτές οι ερωτήσεις τελευταίας στιγμής δεν θα μπορούν να απαντηθούν μέσω τηλεφωνημάτων. Θα πρέπει να πευθυνθούν στον ιστότοπο, εκεί να τα ελέγξει δικηγόρο και όλη αυτή η διαδικασία και δαπανηρή θα είναι και πάρα πολύ χρονοβόρα. Αυτό λοιπόν που θα ζητούσα σε σχέση με αυτούς τους ιστοτόπους είναι να περιμένουμε ένα χρόνο, να δούμε τι θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες εντωμεταξύ. Δεν θα χάσουμε και τίποτα. Και υποπτεύομαι ότι θα δούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείπουν το όλο πείραμα και το εγχείρημα. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να βρούμε μια επαχθή νομοθετική διαδικασία, να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα, οι Αμερικανοί να καταργήσουν εντωμεταξύ αυτή την πρωτοβουλία και εμείς να θέλουμε 10 χρόνια για να το εξαλείψουμε. Θα αυξηθεί πάρα πολύ το κόστο για τι επιχειρήσει μα, θα καθυστερήσει η συγκέντρωση κεφαλαίου και θα πάρουν αλλού αυτά τα κεφάλαια στι χώρε τη Ανατολική Ασία, στην Λατινική Αμερική. Δεν θα μείνει στην Ευρώπη αυτό το κεφάλαιο. Α σκεφτούν πολύ προσεκτικά λοιπόν οι συνάδελφοι για αυτού του ιστοτόπου ε, πριν του ε, θεσπίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φόξ. Πράγματι, οι διαδικασίες που είναι επαχθείς και δαπανηρές, παρόλα αυτά προσφέρουν πλήρη απασχόληση στους ε, δικηγόρους. Ενδιαφέρον λοιπόν αυτό σε επισήμανση. Και τώρα ο κύριος Κλούτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λούλη. Καταρχήν θα ήθελα να σας πενθυμίσω ότι αυτές οι διαμάχες με τις οργανισμούς αξιολόγησης ε, οφείλονται σε κάποια προϊστορία. Με την κρίση είδαμε ότι υπάρχουν προβλήματα μεθοδολογίας και δεν είναι μόνο πολιτικά τα προγράμματα. Γι' αυτό είναι πολύ καλό που συζητάμε το θέμα αυτό και πραγματικά εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας θα ήθελα να πω ότι ουσιαστικά κάνουμε ένα καλό βήμα, ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και καθημερινά θα πρέπει να οδηγούμαστε προς περισσότερη παρακολούθηση και εποπτεία. Το κόμμα μου θεωρεί σαφώς ότι θα πρέπει να υπάρχει μία δημόσια αρχή αξιολόγησης, όμως αυτό βεβαίως δεν είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Η έκθεση του Ζων Πολ βεβαίως πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, γι' αυτό και την ε, χαιρετίζουμε με ικανοποίηση. Το θέμα τώρα του εάν και κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις αν δούμε παραδείγματος χάρη τι έγινε με την Ισπανία, βλέπουμε ότι δεν είναι θέμα ιδιωτικών φορέων ή δημόσιων φορέων και κατά πόσο έχουν δικαίωμα να εκφράσουν την άποψή τους, την αξιολόγησή τους. Το θέμα είναι οι επιπτώσεις, οι οποίες είναι σοβαρότατες και θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, κοινοβουλευτικός έλεγχος και να δούμε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Υπάρχουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές, υπάρχουν τα ελεγκτικά συνέδρια των χωρών και τα συστήματα αυτά, τα ιδρύματα αυτά θα πρέπει να λειτουργούν και να αποτελούν κάποιον, ε, κάποιο αντίβαρο. Διότι καταλαβαίνετε ότι αυτό που συνέβη θα πρέπει να αποφύγουμε να ξαναγίνει και στο μέλλον. Γιατί εδώ αν ξεχνάμε τους δημόσιους φορείς καταλαβαίνετε ότι παρασυρώμαστε σε ένα σύστημα το οποίο έχει σοβαρότατες συνέπειες. Πρέπει να είναι κατά την άποψή μου δημόσιες αυτές οι αρχές, να λειτουργούν με διαφάνεια. Στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει αυτή η διαφάνεια. Υπάρχουν οργανισμοί αξιολόγησης και αν κάποιος θέλει να συνάψει μια συμφωνία, παραδείγματος χάρη με μια άλλη επιχείρηση, μπορεί να ζητήσει μια αξιολόγηση της επιχείρησης με την οποία θέλει να συμβληθεί από έναν ιδιωτικό φορέα. Αυτό δεν μας απασχολεί. Αλλά αν και εδώ θα πρέπει να υπάρχει ποιοτική αξιολόγηση και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα κράτος ε, για το οποίο οι συνέπειες μιας αξιολόγησης είναι εξαιρετικά σοβαρές και έχουν και κοινωνικές πτυχές. Δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που είπαν και άλλοι ομιλητές, αλλά όσον αφορά τις τροπολογίες μας, εδώ φαίνεται ότι δεν ε, θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση για το αν υπάρχει εντολή για μία αξιολόγηση ή δεν υπάρχει εντολή. Πιστεύω δηλαδή ότι το θέμα της πρόθεσης της αξιολόγησης δεν θα πρέπει εδώ να διαφοροποιούν το αν δημοσίως θα δίνονται τα στοιχεία ή όχι. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κλούτε. Οι σκιώδες ηγητές πήραν όλοι το λόγο. Ο κύριος Μπούλμαν έχει ζητήσει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με αυτό που ακούστηκε ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία όσο περισσότερο γίνεται. Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά που δεν έχει γίνει. Αλλά πιστεύω, όπως και ο συνάδελφος Κλούτε, ότι θα πρέπει κάτι να πούμε εδώ για την εξέλιξη αυτής της ε, νομοθεσίας. Τι θα κάνουμε δηλαδή από εδώ και πέρα. Και θυμάμαι τι είχε πει το 2009 ο κύριος Πιτέλα όταν ε, συζητήσαμε πάλι το ίδιο θέμα. Τότε είχαμε πει ότι έπρεπε να ασχοληθούμε με το θέμα που συζητάμε εδώ σήμερα και ακριβώς το θέμα της διάρθρωσης της αγοράς και το θέμα όλων αυτών των φορέων που προσφέρουν υπηρεσίες θα πρέπει να τις συγκεντρώσουμε σε κάποιους φορείς που λειτουργούν βάσει ευρωπαϊκών προτύπων. Είχαμε μιλήσει για το ευρωπαϊκό προφίλ αυτών των οργανισμών. Υπάρχουν πολύ καλά μοντέλα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. εντωμεταξύ καταλαβαίνετε ότι σήμερα δεν είμαστε μόνοι που ζητούμε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι από το ΕΛΚ, ο κύριος Φέρμπερ, άλλοι από τους φιλελεύθερους. Έχω ακούσει απόψεις που συγκλίνουν, ότι κάτι δηλαδή πρέπει να γίνει και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Αλλά θα θέλαμε να επενθυμίσουμε σε όλους τους συναδέλφους ότι η πλειοψηφία ΕΛΚ και Φιλελευθέρων το 2009 είχαν καταψηφίσει αυτό. Και γι' αυτό ακριβώς και στην προηγούμενη θητεία δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε γιατί δεν ε, προχωρήσαμε στην ιδέα να ζητήσουμε από την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω το θέμα αυτό. Χάσαμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία και πολύ θα ήθελα να έχουμε μεγάλη πλειοψηφία σε αυτήν την μελλοντική μας προσπάθεια έτσι ώστε να πάρουμε θέσεις λίγο πιο τολμηρές. Ο κύριος Γκίκολς μίλησε για μια βελτίωση της δομής έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος και υποκτία της αγοράς. Κύριε Μπούλμαν, ξέρετε ότι το ΕΛΚ και οι φιλελεύθεροι εμπνέονται από τον Κόντρατ Άντεναουρ, ο οποίος είχε πει ότι πραγματικά μπορεί κάποιος να αλλάξει άποψη. Ακριβώς αυτό λοιπόν μπορεί να συμβεί και εδώ. Αν κανένας άλλος δεν ζητάει το λόγο, ο κύριος Γκοζές για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ προσεκτικά άκουσα όλους τους συναδέλφους, είχα διαβάσει τις τροπολογίες, άρα δεν με από αυτά που ακούω. Πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να συμπληρώσουμε αυτήν την ρύθμιση. Στο παρελθόν δεν ήμασταν αρκετά τολμηροί. Δεν υπήρχε καμία λύση που να υποστηρίζεται από την πλειοψηφία των μελών. Αλλά το ίδιο πιστεύω θα γίνει και με το θέμα της έκθεσης πρωτοβουλίας όσον αφορά παραδείγματος χάνει τα κρατικά ε, τα κρατικά χρέη. Εδώ πετύχαμε στο Κοινοβούλιο την εποπτεία από την ΕΣΜΑ. Το Συμβούλιο δεν ήθελε. Η Προεδρία δεν ήθελε. Μας έλεγαν ότι δεν ήταν δυνατόν από νομικής απόψεως. Τότε που το ζητήσαμε, όντως δεν ήταν δυνατόν. Χάρη όμως στη στήριξη των συναδέλφων εδώ στην Επιτροπή, καταφέραμε μια νομοθετική πρωτοβουλία με το πακέτο για την εποπτεία και όλοι εμείς γνωρίζουμε ότι η μόνη αρμοδιότητα της ΕΣΜΑ που περιγράφονταν στην πρόταση της Επιτροπής ήταν η εποπτεία, η παρακολούθηση των οργανισμών αξιολόγησης. Μπορούμε λοιπόν τώρα να προχωρήσουμε λίγο. Γι' αυτό και ζητώ να εξεταστεί ξεχωριστά το θέμα της εποπτείας με όλα τα άλλα πολύ σημαντικά θέματα. Να τα αποσυνδέσουμε αυτά Άκουσα λοιπόν πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε. Αύριο με τους Κιώδες θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πνεύμα συνοχής και να υπάρξει πιο σοβαρή ρύθμιση ενός τομέα που έδειξε ότι αν παραμείνει χωρίς κανέναν έλεγχο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά πλήγματα. Έτσι ώστε να μην απομακρυνθούμε από τον αρχικό μας στόχο, γιατί όλοι αυτοί που λένε ότι υπάρχουν πολλοί οργανισμοί αξιολόγησης και η ΕΣΜΑ μόνη της δεν μπορεί να κάνει τίποτα, να μην ε, στηριχτεί από την πλειοψηφία. Κάποιος είπε ότι χρειάζεται βεβαίως ανάθεση κάποιων συγκεκριμένων ε, αποστολών. Ο κεντρικός ρόλος παρόλα αυτά πρέπει να παραμείνει στην ΕΣΜΑ, η οποία είναι η αρχή και για την συντονισμό αλλά και για τις κυρώσεις. Στις 8 Νοεμβρίου λοιπόν θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα των εργασιών μας. Πρόεδρος, ελπίζω η ΕΣΜΑ να έχει και το απαραίτητο προσωπικό για να μπορέσει να διεκπαιρεώσει τις εργασίες της. Θα ήθελα να σας πω ότι αύριο η νομική επιτροπή θα γνωμοδοτήσει επί του θέματος όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Η δεύτερη συζήτηση για τις τροπολογίες θα λάβει χώρα στις 8 Νοεμβρίου και θα ψηφίσουμε στις 9 Νοεμβρίου την έκθεση η οποία θα υποβληθεί στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. Κύριε Ισηγητά, σας εύχομαι καλή συνέχεια. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 18 που είναι η έκθεση του φίλου μου Ντεν Ζαν Έπινγκ, ο οποίος γράφει εξαιρετικά βιβλία για μένα. Πρόκειται για τον ανταγωνισμό, πολιτική ανταγωνισμού 2009. Υπάρχουν επιτροπές που γνωμοδοτούν, ενέργεια, ΙΜΚΟ, βιομηχανία, μεταφορές και τουρισμού. Θα εξετάσουμε λοιπόν τις τροπολογίες. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που είστε τόσο γενναιόδοροι, ώστε να μου δίνετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεισέφεραν στις τροπολογίες, στο σχέδιο έκθεσης για την πολιτική ανταγωνισμού 2009. Κάποιες παρατηρήσεις για τις τροπολογίες, για να ολοκληρωθεί η συζήτηση περί της έκθεσης αυτής. Μέχρι τώρα είχαμε 95 τροπολογίες, οι οποίες ε, ως επιτοπλίστων προσφέρουν ιδιαίτερο περιεχόμενο στην έκθεση. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως μπορούμε να τις ομοδοποιήσουμε ή να τις συγχωνεύσουμε εφόσον είναι παρόμοιες. Υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις που φαίνονται κάπως εκτός θέματος πιστεύω σε μια έκθεση σε σχέση με την πολιτική ανταγωνισμού ή τροπολογίες των οποίων η διατύπωση είναι ασαφής. Εάν η διατύπωση είναι ασαφής και οι παράγραφοι δεν ε, είναι καλά διαρθρωμένε. αρχίζει να μοιάζει με ρωσικό μυθιστόρημα η έκθεσή μας, γιατί όπως ξέρετε τα ρωσικά μυθιστορήματα είναι πάρα πολύ μπερδεμένα. Να αρχίσουμε με τι αιτιολογικέ σκέψει. Συμφωνώ με τι τροπολογίε 1, 5 και 6, καθώ και με τη νέα αιτιολογική σκέψη που προτείνεται στι ε, τροπολογίε 14 ε, και 13, ε, οι οποίε ακολουθούν το πνεύμα του σχεδίου έκθεσή μου και αντιμετωπίζουν συγκεκριμένε ανησυχίες του τροπολογίου. Οι 7 και 8 μου φαίνεται ότι είναι λιγότερο σχετικέ με την έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού, καθώ αφορούν τι αποφάσει για τα δημόσια, για τα δημοσιονομικά ε, ε, και εντάσσονται σε μια ευρύτερη οικονομική συζήτηση. Αυτά είναι θέματα που αφορούν τη δέσμη οικονομικής διακυβέρνησης που συζητούσαμε το πρωί. Και για την ε, τροπολογία 9 του κυρίου Λάμπερτ που μιλά για τι ε, οικονομικές, μακροοικονομικές ανισορροπίε. Και αυτό είναι μέρο τη άλλη δέσμης. Ω προ τι τροπολογίε των παραγράφων πολλέ, αφορούν ε, τίματα του Κοινοβουλίου προ την Επιτροπή να δίνει περισσότερε πληροφορίε ή να διεξαγάγει συγκεκριμένε έρευνε. Αυτέ, μεταξύ των οποίων 15, 16, 19, 29 καθώ και 6 τελευταίε τροπολογίε, τροπολογίες 89-95 νομίζω μπορούν να επαναδιατυπωθούν ώστε να καλύπτουν σχόλια της έκθεσης. Έπειτα υπάρχουν πέντε τροπολογίες που αφορούν τη σταδιακή μείωση του προσωρινού πλαισίου 30 ως 34 όπου αποκλίνουν σαφώς οι απόψεις μεταξύ των μελών της Επιτροπής. Η κυρία Σάγια, για παράδειγμα, μιλά για προσωρινά μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο δυνατόν συντομότερα, ενώ ο κύριος Σφαπ έχει μια τροπολογία η οποία είναι κάπως ασαφής. Λέει ότι μακροπρόθεσμα πρέπει να διακοπούν τέτοια μέτρα. Τελείω. Να πάυσουν. Ιδίω στον τομέα τη αυτοκινητοβιομηχανία. Νομίζω ο κύριο Σβάπ εννοεί ακριβώ το αντίθετο από αυτό που λέει ε, η τροπολογία. Το ιδίω δεδομένη τη κατάσταση τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι ασαφή η διατύπωση των τροπολογιών. Άρα πρέπει να αναζητήσουμε συμβαστικέ λύσεις. Προτείνω να συγχωνευτούν οι τροπολογίες για την στήριξη για τις υπάρξεις παραγράφους καθώς και νέες τροπολογίες 39, 40, 42, 50 με 53. Εδώ το θέμα τέθηκε κατά τη διάρκεια της ακρόασης που οργάνωσε ο κ. Λάμπερτς και είχα και εγώ αυτό το θέμα κατά νου. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσουμε μια συμβαστική τροπολογία, γιατί είναι πολλέ τροπολογίε ακριβώ για το ίδιο θέμα. Και εκφράζουν ακριβώ τον ίδιο φόβο. Στον τομέα τη πολιτική κατά των τραστ, των ομίλων. Εδώ ε, υπάρχουν τέσσερι τροπολογίε μετά την πρόταση τη Επιτροπή. Οι, οι 67 έω 70. Και εδώ θα μπορούσαμε να βρούμε, πιστεύω, συμβαστική λύση προσωπική μου άποψη είναι ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε την ε, τροπολογία 67 της κυρία Σίντφελτ που περιλαμβάνει ένα κατάλογο με εναλλακτικά μέτρα κατά των τραστ των ε, ομίλων και των συγχωνεύσεων. Εδώ λοιπόν το κείμενό της νομίζω ότι είναι καλύτερο και από το δικό μου ακόμη. Είμαι λοιπόν ε, πρόθυμος να το εγκρίνω. Και επίσης υπάρχουν κάποια ζητήματα ίσων ως σημασίας που προκάλεσαν την υποβολή τροπολογιών. 23 και 24 για, την, για τα έσοδα από τον πολιτική ανταγωνισμού. Νομίζω ότι το διατύπωση περιλαμβάνει ήδη το βασικό μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Μπορεί να μείνει ω έχει και δεν χρειάζεται το Ευρωκοινοβούλιο, η Επιτροπή μα να ασχοληθούμε με το ανθρώπινο δυναμικό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ω προ τη στήριξη και τι κρατικέ βοήθειε, νομίζω οι 54, 55, 56, 57 και 58 δεν προσθέτουν τίποτα το ιδιαίτερο, ίσα ίσα είναι κάπως ε, εκτός θέματος. Ε, Παρ' όλα αυτά συμφωνώ με την 55 του κ. Πρεσέντο. Τώρα, οι μισές τροπολογίες που αφορούν την εισαγωγή νέων ε, παραγράφων. Οι 42 και 48 ζητούν από την Επιτροπή να αναλύσει τον αντίκτυπο της κρατικής βοήθειας ε, στις τράπεζες κατά τη διάρκεια των, της κρίσης. Αυτό το ακούσαμε και στην ακρόαση βάσει των τωρινών προτάσεων. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα συμβαστικό κείμενο και σε αυτή την ε, Επιτροπή. Και υπάρχουν πολλές τροπολογίες που αφορούν αφορούν την φορολογική πολιτική. Περισσότερο από ό,τι την πολιτική ανταγωνισμού. Ξέρετε ότι το θέμα αυτό είναι αρκετά ευαίσθητο. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Για αυτόν τον λόγο η προπολογία 27 του κυρίου Λάμπερτ είναι κατά την άποψή μου το καλύτερο σημείο να αναφερθεί η, πολιτική, η, φορολογία, η φορολογική πολιτική και να συνδεθεί με την περιβαλλοντική πολιτική, όπως η πράσινη φορολόγηση. Η, 60, ε, η τροπολογία 60 μπορεί να γίνει αποδεκτή λόγω του υπέρχοντος πλαισίου. Ο ανταγωνισμό στον τομέα τη ενέργεια φαίνεται ότι είναι προτεραιότητα τη πολιτική ατζέντα τη Επιτροπή μα. Υπάρχει και σχέδιο έκθεση τη Επιτροπή η τη κυρία Κοχ Μέριν. Αυτή ε, αυτό το θέμα απεικονίζεται στο σχέδιο έκθεση, όμω κάποιοι θέλησαν να υποβάλουν τροπολογίε ε, σχετικά. Επειδή όμω το ύφο των τροπολογιών του είναι παρόμοιο, είναι κοινό, θα έλεγα να τι συγχωνεύσουμε και να βρούμε μια συμβαστική τροπολογία. Ω προ άλλα θέματα που αναφέρονται λιγότερο συχνά και που έθεξαν συνάδελφοι, όπω για τι υπηρεσίε γενικού οικονομικού ενδιαφέροντο, που είναι πάλι ευαίσθητο θέμα, εκεί θα αναφέρω την 62 του κ. Λάμπερτ. Ε, όπου συνδέει ξεκάθαρα το θέμα αυτό με την πολιτική ανταγωνισμού. Περισσότερο από την τροπολογία του κ. Πρεσέντο που είναι κάπως πιο γενικόλογη. Είμαι υπέρ της τροπολογίας του κ. Πρεσέντο 21 και 22. Και οι δυο τους ε, στηρίζουν την ανάγκη αποκέντρωσης της ε, πολιτικής του ανταγωνισμού κατά των ομίλων συγχωνεύσεων και πιστεύω ότι είναι πιο σημαντική στον τομέα των οικονομικών αυτή η πολιτική παρά στον τομέα των φορολογικών. Και στην ανθρωπολογία σα 66 νομίζω μπορούμε να σταθούμε, ενώ προ τι προτάσει του κ. Λάμπερτ για την 28 μπορώ να συμφωνήσω για την ενίσχυση των προτύπων για το τεχνολογικό κλειδωμά και για τις πιθανές τρευλώσεις του ανταγωνισμού από την τροπολογία 21 και ανάλογα με τις άδειες εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα. Ωστόσο, δεν συμφωνώ την αίτησή σας προς την Επιτροπή να ανασυστήσει την υπηρεσία της. Νομίζω ότι τέτοια υπηρεσία ήδη υπάρχει, άρα είναι περιττή η τροπολογία. Και για την τροπολογία 73, κύριε Λάμπερτ, έχετε υποβάλει πολλέ τροπολογίε και σα ευχαριστώ για αυτό. Το ερώτημα είναι πώ να ορίσουμε την κερδοσκοπία όταν μιλάτε εσεί για την παρακολούθηση των σχετικών αγορών. Πρέπει να προσέξουμε λίγο την ορολογία εδώ. Η κυρία Μακάρθη θέλει να ασχοληθούμε με την ε, τροπολογία 99 για την αγορά με την τροπολογία OTC και ο κύριος Πεσέντο θέλει να εμποδίσει τις, ε, να αλλάξουμε κάτι για τις κινητές αξίες. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς τι είναι με τη διατύπωσή του. Ενώ ο κύριος Πρεσέντο δίνει και πάλι ιδιαίτερη σημασία στον χώρο ενιαίων πληρωμών με τις τοπολογίες 75 και 76 και άλλες. Εδώ χρειάζεται περισσότερη διευκρίνηση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Λίγο πολύ αυτά ήταν τα σχόλιά μου. Νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε συμβαστικέ ε, προτάσει για τα διαφορετικά ε, ζητήματα αυτά και τελικά να καταλήξουμε σε στήριξη τη έκθεση. Σα ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Να δώσω τον λόγο στου σκιώδει εισηγητέ. Ο κύριο Κάριν είναι σκιώδη εισηγητή για το ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον εισηγητή Διάβασα και όλες τις τροπολογίες ε, από τις διάφορες πολιτικές ομάδες και δεν ε, θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Ε, συμφωνώ ότι θα υπάρχουν κάποιες συζητήσεις με τον κύριο Λάμπερτς, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα. Και επίσης να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άντσες Πρεζέ δεν είναι ο εισηγητής των σοσιαλιστών. Ο κύριος Μπούλμαν θα αναλάβει στη θέση του. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, όπως είπατε, ο συνάδελφος Άντσελ Πεδίδο εκπροσωπεί την Επιτροπή μας στην Ινδία, γι' αυτό δεν είναι εδώ. Δεν είναι ότι δεν τον αφορά το θέμα. Ευχαριστώ τον εισηγητή ιδιαίτερα για την παρουσίασή του. Όσον αφορά τις τροπολογίες που έχουμε υποβάλει και που αφορούν τις πιο σημαντικές ιδέες, πρώτον το θέμα του εξυγχρονισμού, του δικαίου ανταγωνισμού που θα πρέπει εδώ να ληφθεί υπόψη για όλους τους τομείς της ενέργειας αλλά και της τεχνολογίας της πληροφορικής και ένα μεγάλο ένας μεγάλος αριθμός τροπολογιών έχουν υποβληθεί γι' αυτό. Ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικό εδώ για την προσθήκη νέων ιδεών. Η θέση μας θα πρέπει εδώ να ενισχυθεί καθότι η σημασία του τομέα αυτού που αφορά τον ανταγωνισμό είναι πάρα πολύ σημαντικός. Κανονισμοί κατά των ε, μονοπωλίων αντιτράστ χρειάζεται γνώση του τι συμβαίνει στον τομέα αυτό, χρειάζεται ανταλλαγή απόψεων και διάλογος και θα συνεχίσουμε αυτές τις συζητήσεις έτσι ώστε να δούμε τι είναι καλύτερο να γίνει και για τη διάσωση των τραπεζών και για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Δεν χρειάζεται περισσότερος ε, περισσότερη στρέβλωση του ανταγωνισμού, γιατί κάθε φορά που υπάρχει τέτοια παρέμβαση ε, αυτός ο ανταγωνισμός υποφέρει. Μιλήσατε για τις υπηρεσίες κοινή ε, Βεβαίως, οι υπηρεσίες αυτές παίζουν ένα, ένα κεντρικό συγγνώμη ρόλο στην αγορά και αυτό αφορά την πολιτική ανταγωνισμού βεβαίως. Είπατε ότι ο συνάδελφος ε, Λάμπερτς αλλά και άλλοι έχουν υποβάλει ενδιαφέρουσες τροπολογίες για το θέμα αυτό και θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά με υποκοδομητικό τρόπο και να βρούμε συμβιβασμό και συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το υποκοδομητικό πνεύμα και δίνω αμέσως το λόγο στην κυρία Ιντβελτ, η οποία είναι η σκιώδη για τους φιλελεύθερους. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και να ζητήσω συγγνώμη και από εσά και από τον εισηγητή για την καθυστέρηση. Αλλά όπω και πολλοί εξημών ε, πρέπει να πηγαίνω από τη μία επιτροπή και τη μία αντιπροσωπεία στην άλλη. Και κάνω ό,τι μπορώ. Θα κάνω μία παρατήρηση πιο γενική διότι είμαι βέβαιη ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να εξετάσουμε πιο προσεκτικά τις τροπολογίες. Κάποιες τις υποστηρίζουμε, κάποιες δεν θα τις υποστηρίξουμε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε ποιος είναι ο σκοπός όλης αυτής της διαδικασίας. Κάθε χρόνο και πέρσι ήμουν εισηγήτρια εγώ για αυτό το θέμα, αλλά κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάει τις απόψεις μας για τις πολιτικές ανταγωνισμού και μετά Έχουμε το χαμόγελο, το συγκαταβατικό του Ευρωπαίου Επιτρόπου, ο οποίος κάθε φορά κάνει το κεφαλιού του. Ε, κάποιοι από εμά ε, μπορεί να υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πολιτική μου ομάδα συνήθω την υποστηρίζει, κάποιοι άλλοι δεν την υποστηρίζουν, αλλά όταν συζητάμε την οικονομική διακυβέρνηση, συζητάμε την αυξημένη συνεργασία, γιατί δίνεται τόσο λίγη πολιτική νομιμότητα στην ε, πολιτική ανταγωνισμού. Και επισημαίνω ότι συνήθω η πολιτική μου ομάδα υποστηρίζει την άγουσα που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει όμως κάποια χώρα, κάποια κυβέρνηση, κάποιο εθνικό κοινοβούλιο που να κάνει οικονομική πολιτική και να μην ε, έχει κάποια επιρροή αυτό στις πολιτικές ανταγωνισμού δεκτό το γεγονός ότι έχουμε συνθήκες, δεν μπορούν να αλλάξουν τα πάντα εν μία νεκτή, κάποιοι δεν επιθυμούν και να τα αλλάξουν. Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης θα πρέπει να είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να παρακολουθήσει στενά τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αν δεν θέλει να ακολουθήσει τις συστάσεις μας, τότε τουλάχιστον θα πρέπει να μας εξηγήσει αναλυτικά γιατί δεν θέλει. Το ζητήσαμε και πέρσι, ο Επίτροπος δεν μας απάντησε και ελπίζω τουλάχιστον φέτος να μας απαντήσει ο Επίτροπος. Ιδάλλως ε, χάνουμε το χρόνο μας εδώ, διότι μπορεί να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση, αλλά αν κάποιος δεν το λάβει υπόψη του, τότε όλη αυτή η διαδικασία είναι μάταιη. Ευχαριστούμε κυρία Ιντφελτ. Η συνθήκη είναι όπως την ξέρετε αλλά ελπίζω ότι το μήνυμά σα θα το ακούσει ο κύριο Αλμούνια και ότι θα ακολουθήσει τις συνετέ σα συμβουλές. Δεν νομίζω όμω ότι υπάρχει κανεί εδώ από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Προσκαλώ λοιπόν τους εκπροσώπους υπεύθυνου για τον ανταγωνισμό να διαβιβάσουν το μήνυμα στον αρμόδιο επίτροπο. Πολύ ωραία. Επόμενος σκιώδης ο κύριος Λάμπερτ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Σόφη τουλάχιστον μας δίνει ε, μια καλή ευκαιρία πρέπει να παραδεχτεί η έκθεση αυτή να έχουμε ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ ενδιαφερόντων ανθρώπων. Ας ε, εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτήν ε, την ευκαιρία. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή για το συστηματικό τρόπο με τον οποίο παρακολούθησε αυτές τις τροπολογίες και για το πόσο ανοιχτόμυαλος φάνηκε. Υποβάλαμε Πολλέ τροπολογίες, πολλοί άριθμε. και έχετε δίκιο ότι δεν είναι όλες ίσως εύστοχες. Ε, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω. Απλώς για το Tax Competition and το Taxation State Aid Unit. Πρέπει να το παρακολουθήσουμε αυτό. Πρέπει να διακρίνουμε εάν χρησιμοποιούμε το σωστό όρο και πού υπάρχει τι μην υποθεί κάτι λάθος. Uh, uh, ε, είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να επιμείνουμε, διότι η φορολογικό ανταγωνισμό είναι κάτι που μα απασχολεί. Να δούμε τη σχετική έκθεση, την έκθεση Μπόντι, διότι είναι πράγματα αυτά που οδηγούν σε δυσλειτουργίε στην εσωτερική αγορά. Και πρέπει πρώτα απ' όλα να βεβαιώσουμε ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα, να δούμε τι αρμόζει εδώ να υποθεί και όχι, αλλά αν μπορεί κάτι να υποθεί να το πει αυτή η έκθεση. Διότι μα ενδιαφέρει μεν το σκέλο του ανταγωνισμού, αλλά και τη φορολογική πολιτική. Είτε πρόκειται για εναρμόνιση είτε όχι. Και θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν στρεβλώνουμε την εσωτερική αγορά. Αυτά είναι τα βασικά μου σχόλια. Κατά τα άλλα, περιμένω θα οργανώσετε συνάντηση των σκιωδών, θα τα δούμε διμερώς, πώς προβλέπετε να διοργανωθείτε. Θα προτείνετε εσείς οι βασικές τροπολογίες, δεν ξέρω τι μέθοδο θα ακολουθήσετε. Ε, ευχαριστούμε. Θα το μάθουμε, μόλις δώσω το λόγο στον ε, εισηγητή και πάλι. Και αφού ακούσουμε όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Έχουμε ακόμη τον σκιώδη εισηγητή της ΚΟΕ, ο οποίος ε, όμως έφυγε. Οπότε να δώσω το λόγο στον κύριο Σβάπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή. Έκανε μια λεπτομερή παρουσίαση όλων των τροπολογιών, μας έδωσε την άποψή του. Εγώ υπέβαλα τροπολογίες που φαίνονται να επικρίνουν το κείμενο, αλλά πιστεύω ότι οι κρατικές ενισχύσεις και όσον αφορά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα ισχύουν, εδώ σαφώς και υπάρχει ημερομηνία καταληκτική. Η τροπολογία 16 που έχει υποβληθεί επίσης με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Κοιτάξτε, το 2008 όταν ήμουν εισηγητής ε, της έκθεσης για τον ανταγωνισμό είχαμε πει ακριβώς το ίδιο με αυτό που λέει αυτή η τροπολογία. Κάθε χρόνο μας ε, απασχολεί το θέμα της ε, πολιτικής ανταγωνισμού με διαφορετικές περιπτώσεις και κάθε φορά η Επιτροπή χρησιμοποιεί σαν επιχειρήματα το τι έγινε το προηγούμενο έτος χωρίς να μπαίνει σε λεπτομέρειες για τις ε, περιπτώσεις. Γι' αυτό και θα ήθελα να ζητήσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για τα ερωτήματα που θέτει το κείμενο αυτό και που δεν έχουν απαντηθεί μέχρι τώρα. Τροπολογία 27, το θέμα της προσαρμογής για την οδηγία 1003. Πρόκειται για την ανάγκη μεταρρύθμισης και εδώ θα πρέπει η Επιτροπή είτε να υπερψηφίσει, είτε να υποστηρίξει μάλλον, είτε να απορρίψει. Αυτό όμως δεν έγινε μέχρι τώρα. Η μεταρρύθμιση αυτή ε, βεβαίως που αφορά το θέμα του ανταγωνισμού δεν έλαβε χώρα. Το 2003 είχαμε φτάσει σε έναν συμβιβασμό και τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, η Επιτροπή θεώρησε τότε, μας άφησε να εννοήσουμε ότι υπάρχει δυνατότητα για μια ευρύτερη ερμηνεία αυτής της οδηγίας, ότι είναι αρμόδια τα κράτη-μέλη με την Επιτροπή και ότι σαφώς και χρειάζεται μια μεταρρύθμιση, υπάρχει ανάγκη μεταρρύθμισης. Επιγόντως θα έλεγα εγώ, τότε ο Επίτροπος, ε, αν θυμάστε στην ακρόαση εδώ στην ε, Επιτροπή μας μίλησε για τις επιχειρήσεις ε, μόνο product businesses, για τις επιχειρήσεις αυτές που έχουν ένα μόνο ε, αντικείμενο, λέγοντας ότι θα τύχουν ειδική μεταχείριση Επίσης, όσον αφορά τις κυρώσεις, ε, τις χρηματικές, τα χρηματικά πρόστιμα, όπως είχε συζητηθεί τότε, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και σε αυτήν την πρόταση. Και με αυτόν τον τρόπο θα πιέσουμε την Επιτροπή να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά που ακόμα δεν έχει απαντήσει. Πρόεδρος, κανένας δεν έχει ζητήσει το λόγο. Κυρία Ίνβελτ, υπάρχει εκπρόσωπος της Επιτροπής. Αν θέλετε να επαναλάβετε την ερώτησή σας, η κυρία Χάμιλτον είναι παρούσα και κανείς άλλος δεν ζητάει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα βέβαια να παρέμβω στο ρόλο του εισηγητή. Η ερώτησή μου είναι απλή. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε θέματα πολιτικής ανταγωνισμού, θεωρώ, όπως είπα και νωρίτερα, ότι όταν συζητάμε θέματα οικονομικής διακυβέρνησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ανταγωνισμός είναι αναπόσπαστο τμήμα της οικονομικής διακυβέρνησης και παρά το γεγονός ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τουλάχιστον ηθική υποχρέωση προς τους Ευρωπαίους πολίτες να απαντήσει αναλυτικά σε όλες τις ερωτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν έγινε κάτι τέτοιο πέρσι, όπως επεσήμανε και ο συνάδελφος ο κ. Σβάμπ, και θα θέλαμε τουλάχιστον φέτος ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί τις συστάσεις μας και αν ε, δεν τις λάβει υπόψη της να μας πει τουλάχιστον για ποιο λόγο. Δεν ξέρω αν η κυρία Χάμιλτον θέλει να απαντήσει. αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να διαβάσει το μήνυμα στον Επίτροπό τη. Θέλετε να απαντήσετε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Απλώ να πω ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα ε, φέτος για να απαντήσουμε τι ερωτήσει. σα. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή τώρα. Έχετε πολλά πράγματα να μας πείτε, διότι πρέπει να καταλήξετε σε πολλές συμβαστικές τροπολογίες. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ελπίζω να είναι βανάγνωστα και κατανοητά. Θα ψηφίσουμε στις 30 Νοεμβρίου, επομένως έχετε χρόνο. Και επειδή δεν έχουμε προβλέψει δεύτερη συζήτηση για τις τροπολογίες, σίγουρα θα είστε διαθέσιμος να οργανώσετε μια συνεδρίαση με τους κοιόδη εισηγητές, ώστε να μπορέσετε να μας βοηθήσετε να ψηφίσουμε καλύτερα στην Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την παραστήριση του κυρίου Μπούλμαν εξ του ονόματος κυρία Σάντσες Πρεσέδο. Σαφώς τα θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος είναι πολύ σημαντικά, αλλά μας ενδιαφέρει και η σωστή διατύπωση. Υπάρχει ανάλογη τροπολογία του κυρίου Λάμπερτς, και νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα ακριβές κείμενο το οποίο θα είναι ευανάγνωστο. Όσο πιο μακροσκελές είναι τόσο πιο ε, αμφίσιμο γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε λίγο τη διατύπωση της τροπολογίας. Κυρία Ίνεντβελτ, ε, όταν δεν ήσασταν εδώ στην αίθουσα, ε, σας συνεχάριν για την ε, τροπολογία 67. Είπα ότι είναι καλύτερο το δικό σας κείμενο από το δικό μου, επομένως ε, θα δεκτώ την τροπολογία σας και θα δω και τα θέματα τα οποία ανέφερε ο κύριος Φαμπ. Ε, όπου χρειάζεται περαιτέρω δουλειά και μελέτη για θέματα τα οποία έχουν ξανασυζητηθεί. Ώστε όλα να έχουν μια πραγματική σημασία. Επίσης, Είχα ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν υπάρχει μια text unit ή όχι, αλλά μου είπαν ότι υπάρχει ε, και αποτελείται από πολύ λίγους ανθρώπους. Δεν ξέρω, μπορεί να πίνουν καφέ και να διαβάζουν εφημερίδες, οπότε να μην κάνουν πολλή δουλειά. Θα πρέπει να ανακαλύψουμε αν υπάρχει τέτοιο τμήμα και αν λειτουργεί. Κύριε Σβάμπ, για την τροπολογία που ρωτήσατε, ε, μπορεί να είναι θέμα μετάφρασης, διότι εγώ είδα την αγγλική μετάφραση και εκεί λέει in the long term, μακροπρόθεσμα και το ότι θα πρέπει να σταματούν τα μέτρα στα πλαίσια του προσωρινού πλαισίου. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι προσωρινό και θα πρέπει κάποια στιγμή να διακοπεί. Είστε μέλος του ΕΛΚ και η κυρία Σάγια είπε ότι θα πρέπει να σταματήσει το συντομότερο δυνατόν. Δεν ξέρω πότε είναι αυτό το συντομότερο δυνατόν, αλλά θα πρέπει να σταματήσει γιατί στρεβλώνει τον ανταγωνισμό αν συνεχιστεί κάτι τέτοιο. Και τέλος, ως προς τη διαδικασία θα ήθελα να συναντηθώ με τους κοιόδης εισηγητές ώστε να εντοπίσουμε τα θέματα στα οποία θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό και στη συνέχεια θα κάνω μία απόπειρα να ετοιμάσω κάποιο συμβιβαστικό κείμενο, θα ξανασυναντηθούμε, θα δούμε την ακριβή διατύπωση και ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου. Κατά τα λοιπά, κυρία Πρόεδρε, το μασάζ του Επιτρόπου θα τα αφήσω στην κυρία Ίνετβιλτ. Est-ce que Madame la représentante de la Commission veut répondre à cette question Ναι, θα σας απαντήσει η Κοιτάξτε, θα δούμε βεβαίως πώς θα ρυθμιστεί το θέμα του τι κάνουν οι μεν και οι δε. Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει μια τέτοια υπηρεσία η οποία δεν ασχολείται μόνο για το θέμα αυτό. Ασχολείται κυρίως με το φορολογικό θέμα, αλλά όχι μόνο. Σαφώς διαβάσατε και στον τύπο διάφορες ενισχύσεις οι οποίες παρέχονται στα κράτη-μέλη και η υπηρεσία αυτή εργάζεται. Αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχει, η Επιτροπή εξετάζει όλες τις ενισχύσεις οποιασδήποτε μορφής. Λοιπόν, άρα θα μου δώσετε και εμένα κάποιες διευκρινήσεις. Ακόμα και αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία. Πρόκειται για θέματα εξαιρετικά περίπλοκα και μπορεί να είστε αποτελεσματικοί μόνο και εφόσον καλύπτεται όλη την τεχνική γνώση εμπειρογνωμοσύνη σε ένα σημείο συγκεκριμένο. Πόσα άτομα εργάζονται λοιπόν για τα φορολογικά θέματα. Γιατί λέτε δεν εργάζονται μόνο. Πόσα είναι και πόσο χρόνο από τον χρόνο εργασία τους δαπανούν για το θέμα αυτό της φορολογίας. Θέλετε να απαντήσετε κυρία Μπρόμς ή θα απαντήσετε αργότερα γραπτός. Ναι, επειδή μου ζητάτε λεπτομερή απάντηση θα το κάνω γραπτός. Τα άτομα που ασχολούνται με τις ε, ενισχύσεις ε, ασχολούνται μόνο με αυτό, αποκλειστικά και μόνο. Και πρόκειται για ειδικού του δημοσιονομικού τομέα δεν είναι τόσο πολύ πολυδιάστατη κύριε Λάμπερτς όπως είμαστε εμείς. Τελείωσε η συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου. Θα υποβληθούν φαντάζομαι συμβιβαστικές τροπολογίες. Πολύ προσωπικά θα ήθελα να εκφράσω μια επιθυμία. Καλό θα ήταν αν οι τροπολογίες οι συμβιβαστικές δεν ε, μας υποβληθούν την προηγούμενη το βράδυ στις 9 όπως έγινε για την έκθεση Φεγιό. Γιατί δεν είναι ευχάριστο να έχουμε τις τροπολογίες τελευταία στιγμή έτσι ώστε τα απλά κακόμοιρα μέλη σαν και μένα να μπορούν να τις διαβάσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι τα διάφορα. Όμως δεν επιμένω, αφού δεν υπάρχουν. Αν έχετε όμως κάτι να πείτε βεβαίως, δεν βλέπω κανέναν. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα 8 Νοεμβρίου, Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου στις 3 και 9 Νοεμβρίου το πρωί και το απόγευμα. Τέλος της συνεδρίασης.